Καλημέρα σε όλους σας. Θα σας παρακαλούσα να καθίσετε. And, uh, welcome you to the meeting. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε παρτία τώρα για να μπορέσουμε να συνεδριάσουμε. Σας καλωσορίζω. Καλημέρα σας και πάλι και κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασής μας για σήμερα. Θέμα πρώτον. Έγκριση της σημερινής διάταξης. Μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ορίστε Βανίστεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μπορούμε. Yes, we can. And addition, yesterday we did. Εκτός αυτού, εχθές το βράδυ δεν συνεδριάσαμε, ε, γιατί δεν είχαμε θέματα στη μέση διάταξη χθες το απόγευμα. Σήμερα έχουμε μόνο μελέτες. Ε, στις ανακοινώσεις ε, της Προέδρου θα είχα μία πρόταση εγώ για να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια για ορισμένα θέματα. Θέλετε να το πω τώρα ή όταν ε, έρθει το σημείο 3 στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου, ό,τι πείτε εσείς Πρόεδρε. Thank you. Thank you very much. right. We didn't... Ναι, ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Χθε δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, αλλά θα έχουμε συνεδρία συντονιστών σήμερα. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε και αυτή την απόφαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών για την πρόταση που έχετε αυτή που μας είπατε για την προφορική σας ερώτηση. Συμφωνείτε? Ο κύριος Βανίστε Ρόι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα τώρα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε στους συντονιστές αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ε, ακριβώς επειδή είχαμε χτες χρόνο για να εργαστούμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δουλεύουμε και όχι να περιμένουμε. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία εδώ για τις πιθανές καθυστερήσεις πολλών προγραμμάτων. Το 2014, ας πούμε, αν προσπαθήσουμε να το δούμε στην περίοδο 2014-2020 είναι μόνο περίοδος προγραμματισμού, δεν έχει αρχίσει ουσιαστική δουλειά. Και το 2015 θα υπάρξει κατακλυσμός πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία σε πρόγραμμα. Όλο συζητάμε ε, για δημιουργία θέσεων ε, εργασίας, για ε, επενδύσεις και που τι κάνουμε εμείς για τη συνοχή στην Ένωση. Και αν το δούμε και βαθύτερα, έχουμε τους στόχους για την οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η φορεία, ε, ηλεκτρονικά και άλλα, η τεχνολογία της πληροφορίας. Και βεβαίως έχουμε και το πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών, εκτός αυτού. Λοιπόν, πολιτικά μπορεί να ήταν ευφυές όχι απλώ να καθόμαστε εδώ και να τα καταλαβαίνουμε μόνοι μα όλα αυτά, αλλά να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα και να ζητήσουμε ήδη ε, το Νοέμβριο στην Ολομέλεια να μα παρουσιάσουν την κατάσταση των πραγμάτων. Όπω είπατε μπορούμε να κάνουμε ένα τώρα μεγάλο συνολικό κείμενο με τέσσερι ερωτήσει που θα είναι ωραίο και σοφό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει όλοι από όλες τις πολιτικές ομάδες και να το στείλουμε τώρα από τη γραμματεία. Χθε μίλησα με την Κωνσταντσα Κρέλ για αυτό το θέμα. Το έχουμε κοιτάξει δηλαδή ε, αυτό το κείμενο τις ώρες που είχαμε προγραμματίσει για συνεδρίαση της Επιτροπής. Αν θέλετε να το δείτε όλοι και αν μπορούμε να το αποφασίσουμε, μπορούμε να το κάνουμε ε, προφορική ερώτηση της Επιτροπής. Ε, ή μπορείτε να το κάνετε μέσα των πολιτικών ομάδων από τους συντονιστές. Το θέμα δεν είναι πώς θα γίνει, αλλά θέλουμε να, να, να το συζητούμε πολιτικά, όχι διαδικαστικά όλο αυτό για τον έλεγχο κτλ. Συμφωνώ απολύτως. Να το στείλουμε και κοιτώ τώρα τους συντονιστές, τα μέλη και τους βοηθούς να βγει σήμερα η ερώτηση, όχι να περιμένουμε μέχρι την επόμενη ε, συνεδρία των συντονιστών, γιατί θα καταλήξουμε κάπου το 15 στην Ολομέλεια, ενώ μιλάμε για το 14. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η Πρόεδρος. Αυτό το χαρτί που μου δώσατε τώρα φωτοτυπείτε. Ε, σας ευχαριστώ. είχε θα λάβουν όλοι ένα αντίγραφο και κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης των συντονιστών θα πάρουμε απόφαση. Σας καλύπτει αυτό κύριε Βανίστερο, είστε εντάξει. Ναι, ναι, βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Άλλες προτάσεις για την ημερήσια διάταξη σήμερα. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Το δεύτερο σημείο είναι η άγκριση των πρακτικών. Έχουμε τα πρακτικά ε, των εξης συνεδριασεων συνεδριάσεων 22-23 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου και 6 Οκτωβρίου. Τα έχετε στα χέρια σας, το σχέδιο των πρακτικών. Όσοι ήθιστε, αν δεν έχετε καμιά αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Διαφωνεί κανείς. Όχι. Ή έχετε να προβάλλετε καμία ένσταση για τα πρακτικά. Ωραία. Θα εγκριθούν όπως είπαμε. Ανακοίνωση, του Πρόεδρου. Σημείο 3. Δεν έχω... Δεν σας κάνω ανακοίνωση. Το τέταρτο θέμα είναι το πρώτο ουσιαστικό θέμα σήμερα το πρωί μια μελέτη για να συζητήσουμε τα ευρήματά της με θέμα την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, της προετοιμασίας και τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών. Ζητήθηκε από την Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο του 2013 πέρυσι, η ε, μονάδα έρευνας που υποστηρίζει ε, το τμήμα πολιτικής ε, Β ζήτησε από μια εταιρεία στη Βιέννη, Μέτρης, με την οποία έχουμε σύμβαση πλαίσιο να ε, διεξάγει τη μελέτη με στόχο να μελετήσουμε τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών για να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχή στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και να δούμε πώς έχει προετοιμαστεί η κάθε διοίκηση για να αρχίσει σωστά η προγραμματική περίοδος. 14 περιπτώσεις μελετήθηκαν και αναλύθηκαν και θα μας τα παρουσιάσει όλα αυτά η κυρία Χριστίν Χάμζα που παρευρίσκεται και είναι κύρια σύμβουλος στην εταιρεία ΜΕΤΗΣ. Μετά την παρουσίαση θα δώσω το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις και προτάσεις. Παρακαλώ, κυρία Χάμζα, έχετε το λόγο. <coughs> Thank Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να παρουσιάσω μία μελέτη που ήταν ε, ιδιαίτερα, που αποτελούσε μάλλον πρόκληση και ήταν και χρονοβόρα. Μας απασχόλησε για 10 μήνες κατά την καυτή φάση της περίοδου προγραμματισμού που δεν έχει λήξει ακόμα. Άρα υπάρχει στάτους κουβό, υπήρχε δηλαδή, κατά τη διάρκεια της αποτίμησης. Θα ήθελα να σας πω πώς ε, επιλέξαμε τα κράτη-μέλη για τις κατά περίπτωση μελέτες και να σας μιλήσω και για τις προκλήσεις ε, της ε, εταιρικής συμφωνίας πριν μιλήσω για θέματα ικανότητας και για τις συστάσεις. Η επιλογή των κρατών μελών για τις ε, κατά περίπτωση μελέτες είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί μέσα στα πλαίσια της συνολικής τάσης των κρατών μελών, άρα λάβαμε υπόψη διάφορες ε, παραμέτρους, δηλαδή λάβαμε υπόψη το κριτήριο ε15 και ε12 ε συν 1, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα μεγέθη των ε, διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και τα μικρά. Και ορισμένα κράτη-μέλη είδαμε ότι δεν άλλαξαν τη διάρθρωση και τα ποσά των προγραμμάτων, ενώ άλλα μίλησαν τα επιχειρησιακά προγράμματα και έλαβαν υπόψη τις δυνατότητες των ε, ταμείων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ. Άρα επιλέξαμε 14 χώρες, την Αυστρία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο και Σουηδία, με μικρό προϋπολογισμό Ιταλία, ε, Ελλάδα ε, και την Γερμανία, καθώς και τη Γαλλία που είναι μεγάλες ε, χώρες εκτός, ε, ως προς τη χρήση αυτών των κονδυλίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνένα ε, Εστονία, ε, Κροατία και Βουλγαρία. Επιλέξαμε την Κροατία γιατί πρόκειται για μια νέα χώρα και μας ενδιαφέρει το πώς ε, εργάζεται και χρησιμοποιεί τα διαρθρωτικά ταμεία. Και επίσης την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Αυτό που μας ε, απασχόλησε είναι να δούμε τα, τις δυσκολίες των εταιρικών συμφωνίων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τώρα καταγράφουμε τις δυσκολίες γιατί με βάση αυτές ε, ορίζουμε και τις συστάσεις μας, άρα δεν είναι όλα τα στοιχεία αρνητικά ως προς την ε, διοικητική ικανότητα της εφαρμογής του προγράμματος προσπαθήσαμε να αποτιμήσουμε το ζήτημα και να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε αυτή την πληροφορία καθώς ε, και την προετοιμασία των ε, διαχειριστικών αρχών και των φορέων εφαρμογής έτσι ώστε να προβούμε σε συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως προς τα θέματα προκλήσεων στις συμφωνίες εταιρική σχέσης, θα ήθελα να πω ότι έγιναν πολλές αποτιμήσεις εξ άντε και είδα ότι υπάρχουν και θέματα επικοινωνίας. Η επικοινωνία όμως αυξήθηκε μεταξύ διαφόρων τμήματων και υπήρχε θετικό input των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, διότι προγενέστερα τα διάφορα τμήματα δεν συζητούσαν το θέμα της εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων. Γιατί υπήρχαν ζητήματα αρχής. Από την άλλη πλευρά όμως η προσαρμογή των ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, δεν λειτουργήσαν σε όλες τις χώρες, δηλαδή αυτή τη στιγμή ορίζονται και αποτιμούνται, αλλά δεν υπήρξε πραγματική προσαρμογή από πλευράς ε, χρόνου και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα σε εκείνες με μικρό προϋπολογισμό και ένα πρόγραμμα ΕΤΠΑ, θεωρήσαμε ότι η εταιρική σχέση ίσως ε, αποτέλεσε επικάλυψη. Αυτό δεν ισχύει, αλλά αυτή την εντύπωση είχαν σε ορισμένες χώρες όπου η μακροοικονομική κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, ε, ήταν δύσκολο να έχουμε μία θεματική ενότητα, διότι όλοι ήθελαν να γίνει ένας επιμερισμός των κονδυλίων. Επίσης, οι κυβερνητικές αλλαγές, οι εκλογές, η διενέργεια εκλογών ήταν ε, ζήτημα για την Ουγγαρία, για την Ιταλία, επί παραδείγματι και στη συνέχεια υπήρχαν πολιτικές, μάλλον δεν υπήρχαν πολιτικές δεσμεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Και ενώ υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών φορέων, υπάρχει δυνατότητα για βελτίωση. Τώρα, ποιες θα οι δυσκολίες των, ε, της επιχειρησιακής ανάπτυξης. Α, ε, πρόκειτο για την επιλογή θεμάτων. Δηλαδή όλα τα τμήματα συμμετείχαν σε αυτή τη συλλογιστική για να δούμε πόσο περισσότερα κονδύλια ε, μπορούσαν να λάβουν από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά εδώ Είχαμε να κάνουμε και με περιφέρειες που είχαν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ορισμένε ε, χώρες δεν ήθελαν να αλλάξουν το επιχειρησιακό περιεχόμενο, δηλαδή προϋπήρχε γιατί έπρεπε να αλλάξει, θεώρησαν. Και υπήρξαν και πολλές διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Δηλαδή ως προς την ερμηνεία των ε, δικτών και αυτό ήταν ε, κάτι το ιδιαίτερο, το ιδιαίτερα χρονοβόρο. Ε, μεταξύ περιφερειακού, τοπικού και εθνικού επίπεδου. Και στη συνέχεια ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι ορισμένα κράτη-μέλη άρχισαν την διαδικασία προγραμματισμού πολύ νωρίς, διότι το υλικό καθοδήγησης δεν ήταν έτοιμο και χρειάστηκε να γίνει επαναπρογραμματισμός με βάση το ε, υλικό αυτό που άλλαξε σε σχέση με τον προγραμματισμό δηλαδή και τις κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα, ως προς τα θέματα ικανότητας, είχαμε διάφορες πηγές, γιατί οι συνεντεύξεις με τα κράτη-μέλη και τη δημόσια διοίκηση δεν επαρκούσε για να υπάρξει ευρεία ε, κατανόηση του ζητήματος. Γι' αυτό είχαμε τα έγγραφα αρχής, τα βασικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διευθύνσης ε, Ρέγγιο. Επίσης, ο εξάντε προγραμματισμός μας και βεβαίως υπήρχαν, έγιναν και συνεντεύξεις με την διαχειριστική αρχή. Έχουμε εννέα ζητήματα, μείζωνα ζητήματα που αφορούν την ικανότητα, ότι δεν υπάρχει στρατηγική προσέγγιση, υπάρχει ανεπαρκής ε, προγραμματισμός, ε, δεν υπάρχει λογοδοσία, ε, υπάρχει ε, ανεπαρκής δημοσιονομικός έλεγχος και ανεπαρκής, ανεπαρκής διαχωρισμός μεταξύ των πολιτικών επιλογών και της δημόσιας διοίκησης σε ζητήματα καταβολής πληρωμών. Επίσης, δεν υπάρχουν επαρκείς δεξιότητες και εξοπλισμός. Αυτό ισχύει στις περισσότερες χώρες, σε όλες τις χώρες, αλλά Υπάρχει ανεπαρκής προγραμματισμός, ε, ε, αλλαγή στο προσωπικό και ανεπαρκής δεξιότητες, καθώς και συντονισμός ο οποίος εκλείπει. Γι' αυτό επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε αυτά τα τέσσερα ζητήματα έγινε μία ε, αυτοαποτίμηση και οι διαχειριστικές αρχές ε, σε αυτή την αυτοαποτίμηση έδωσαν, έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα με αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αρχικό της έγγραφο. Άρα η διοικητική ικανότητα που καλύπτεται στο, στην θεματική ενότητα 11 όπου υποστηρίζονται τα ημίμια ΜΜΕ, ε, εδώ υπάρχουν οι μεγαλύτερες λήψεις και το λιγότερο αποτελεσματικό είναι οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν το περιβάλλον και τις υποδομές. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό, διότι τα σχέδια υποδομής είναι πιο χρονοβόρα, πολυσχηδή και με πολλά διοικητικά ζητήματα και προγενέστερο προγραμματισμό και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ε, σαφής γνώση και πραγματογνωμοσύνη. Άρα το βασικό βασικό ζήτημα στις συνεντεύξεις ήταν η έλλειψη πόρων, γνώσης και πείρας του νέου προσωπικού, διότι αλλάζει συνεχώς το προσωπικό. Αυτό το θέμα αφορά τα κράτη-μέλη όπου οι πληρωμές δεν ήταν τόσο προβληματικές. Αυτό είναι ένα βασικό λοιπόν ζήτημα. Ένα άλλο θέμα ήταν η επικάλυψη της, του προγραμματισμού, της διαχείρισης του προγραμματισμού 713 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε πλέον αυτό το πρόγραμμα, το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που μας απασχόλησε και στην προγενέστερη περίοδο, 7-13. Δηλαδή είχαμε δύο περιόδους προγραμματισμού, παράλληλες ε, περιόδους προγραμματισμού. Στη συνέχεια, από τις συνεντεύξεις και από τις μελέτες, ε, και από τις έρευνές μας στα γραφεία είδαμε ότι υπάρχουν ζητήματα ικανότητας, ιδιαίτερα χώρες που έχουν ομοσπονδιακό χαρακτήρα ή ισχυρές περιφέρειες που έχουν πιο ε, συγκεντρωτικό χαρακτήρα λήψης αποφάσεων. Κάτι το οποίο ε, διονγκώνει το θέμα της, ε, του συντονισμού. Δηλαδή στην Αυστρία υπάρχει ένα κεντρικό πρόγραμμα, αλλά δεν σημαίνει ότι οι περιφερειακές αρχές δεν αποτελούν βασική διοίκηση και ασχολούνται με θέματα διαχείρισης και χρηματοδότησης μέσα στα πλαίσια του ομοσπονδιακού χαρακτήρα αυτής της αντίληψης δηλαδή που επικρατεί. Επίσης υπάρχει ε, ανεπαρκής εκδήλωση ενδιαφέροντας, Δηλαδή δεν υπάρχει επαγγελματισμός και οι δικαιούχοι δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δεν υπάρχει το σωστό χρονικό πλαίσιο και στη συνέχεια υπάρχουν προβλήματα στην αποτίμηση των προγραμμάτων. Αυτό το βίωσα και η ίδια, γιατί βλέπω ότι πολλά προγράμματα είναι πολύ καλά στην αρχή, αλλά αν σκάψετε λίγο κάτω από την επιφάνεια και αν έχετε πείρα, κατανοείτε ότι η περιγραφή τους δεν είναι επαρκής. Επίσης ε, υπάρχει θέμα αποτίμησης και διασάφησης των ρόλων και το θέμα της επικοινωνίας αφορά και τους δικαιούχους ε, μεταξύ τους αλλά και διάφορα τμήματα και διάφορα επίπεδα, δηλαδή εθνικό και περιφερειακό. Στη συνέχεια, ε, δυστυχώς, οι δικαιούχοι δεν είναι σε θέση πάντα να θέσουν σε εφαρμογή τα προγράμματα. Έχουν γίνει πολλές ε, προτάσεις βελτίωσης, δηλαδή ζητήματα όπου τα κράτη-μέλη προτείνουν βελτιώσεις και οι περισσότερες αναφέρονται στα επιχειρησιακά προγράμματα. Και πολλές αφορούν την εξάντε ερεσιμότητα. Δηλαδή σε ορισμένες χώρες γίνονται νομικές ε, προσαρμογές, οι κατάλληλες νομικές ε, προσαρμογές για να ανταποκριθούν στα διαρθρωτικά ταμεία, έτσι ώστε να εφαρμόζονται καλύτερα. Και η εναρμόνιση των κανόνων των διαρθρωτικών ταμείων με τους εθνικούς κανόνες. Άλλες χώρες ανέφεραν ότι προτίθενται να αποδώσουν ε, ε, σαφέστερες ε, αρμοδιότητες και ευθύνες, δεν αναφέρεται πώς και άλλες χώρες έχουν μειώσει τον αριθμό των εφαρμοστικών αρχών, όπως η Εσθονία. Επίσης, έχει σημασία η ολοκλήρωση των ε, ευρωπαϊκών και εγχωρίων προγραμμάτων. Η Πολωνία ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην προσαρμογή στα, ε, στους κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων με τους εθνικούς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 Επίσης, χρειάζεται μια καλύτερη στοχοθέτηση στην επιλογή προγραμμάτων και αυτό ε, αφορά θέματα συνοχής που ανέφεραν όλοι. Δεν ξέρουμε βεβαίως πώς θα εφαρμοστεί αυτό το θέμα του οικοχίζων. και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει σαφής ε, ουσιαστική ε, εφαρμογή. Επίσης, ενίσχυση του, της επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης. Δεν ξέρουμε πώς θα επιτελεστεί αυτό. Ελπίζουμε να το δούμε στην ε, εκ των προτέρων ε, αιρεσιμότητα. Στη συνέχεια ε, μας απασχολεί η υποστήριξη της ανάπτυξης ικανότητας μεταξύ των μικρών τοπικών φορέων, όπως ισχύει στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Τα συμπεράσματα σε σχέση με τα θέματα ικανότητας, αν μπορούμε να τα εντάξουμε σε μία διαφάνεια, έχουν ως εξής. Υπάρχει σωρία προβλημάτων, αλλά οπωσδήποτε έχουμε αποκτήσει πείρα από την προγενέστερη περίοδο και από τις συνεντεύξεις είδαμε πως οι διαχειριστικές αρχές αντέδρασαν στα δικά μας ε, ζητήματα και αυτό αποτελεί μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο προγραμματισμού. Έχουμε μείωση προγραμμάτων και τη συγκέντρωση των διοικητικών ε, ζητημάτων και αρμοδιοτήτων. Αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη βελτίωση, όμως η σαφής ή, ή μάλλον η μαλλον η συγκεκριμενη ο συγκεκριμένος προγραμματισμός και εφαρμογή της διαχείρισης δημιουργεί προβλήματα, διότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά τμήματα που ασχολούνται με τα διαρθρωτικά ταμεία ανάλογα με το ποιο πρόκειται. Επίσης, ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα συγκεντρωτισμού και συγκέντρωσης περισσότερο των ε, διοικητικών ε, διαχειριστικών αρχών. Γι' αυτό αντιμετωπίσαμε και θέματα εφαρμογής στην προγενέστερη περίοδο προγραμματισμού. Και οι εθνικές και περιφερειακές ε, διοικήσεις δεν έχουν προσαρμοστεί ε, με τις διοικήσεις των διαρθρωτικών ταμείων. Άρα, ποιες είναι οι συστάσεις. Προτείνουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε καταρχήν τις εξάντε ερεσιμότητες. Έχουμε μέχρι το 16 για την εφαρμογή αυτών των ε, εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων που δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί και εδώ χρειάζεται παρατήρηση και εδώ υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία με, την ε, ευρωπαϊκή, με τα ευρωπαϊκά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη εικόνα για την πρόοδο των συγκεκριμένων σχεδίων. Για να δούμε τι συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, τμήματα ε, που ασχολούνται με την διοικητική ικανότητα, όπως ε, ακριβώς προείπα. Τέλος. Γενικότερα θα πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Χρειάζεται τυποποίηση των προγραμμάτων και από τα δύο θεσμικά όργανα μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού της Επιτροπής και του ελέγχου της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χρειάζεται μια επιτάχυση του μελλοντικού προγραμματισμού των ε, διαφόρων φάσεων του 2020+. Καλύτερη προσαρμογή πληροφόρησης μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου, και τέλος, ε, καλύτερη γνώση σε σχέση με τις δυνατότητες των διοικήσεων και της διοικητικής ικανότητας. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις διοικητικές ικανότητες και χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί ε, μία ε, μικρή παρουσίαση των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, προσοχή σας και θα ήθελα να μου υποβάλλετε ερωτήσεις. And, uh, Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Έχουμε όλη τη μελέτη βεβαίως και τα παραρτήματά της. Είναι εντυπωσιακό το έγγραφο. Θα δώσω το λόγο τώρα στα μέλη της Επιτροπής, ερωτήσεις και προτάσεις. Ο κύριο Βανίστερ Ρόι. Σίκο και οι λοιποί θα ακολουθήσουν ε, κατάλογο ως αγορητών. Ο κύριο Φανίστερ ε, Ρόι. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Ολλανδικά. Στην αρχή της περίοδου αυτής της προγραμματικής είναι καλό να μελετούμε πάρα πολύ σοβαρά και προσεκτικά τις ε, μελέτες ε, που κυκλοφορούν για να δούμε αν συνάδει η πρακτική με τη θεωρία των προγραμμάτων. Έχουμε διάφορα παραδείγματα που χρειάζονται προσοχή. Έχω πολλές ερωτήσεις, μερικές δηλαδή. Ψάχνω λίγο τη μέθοδο με την οποία μετρήσατε. Το ξέρω ότι είναι ποιοτική βέβαια η μελέτη, αλλά καμιά φορά θα πρέπει να μελετάτε αν είναι αρκετή έτσι, αυτή η διοικητική ικανότητα. Αν ρωτήσει κάποιον χασάπι είναι καλό το κρέα σου, θα σου πει καλό είναι. Άμα πάτε όμως να, ρωτήσετε επίσης ε, ε, τις ελεκτικές αρχές ή τις ε, θα σου πούνε μια χαρά τα πάμε. Δεν ρωτάς τον ενδιαφερόμενο που, που κρίνεται, τον ελέγχεις. Έχετε συζητήσει λοιπόν με εκείνους που στις πόλεις, περιφέρειες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, σχολεία ε, έχουν ε, μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό ήταν το πνεύμα στην αρχή που μας ενέπνευσε για τον κώδικα συμπεριφοράς και διοντολογίας. Για το πώς θα δουλεύουν τα κράτη-μέλη. Ε, σαν να ίσχυε ε, ήδη ο κανονισμός με εταιρική σχέση, με συνεργασία στη βάση. Λοιπόν, εγώ ψάχνω τη μέθοδο, γιατί στην πολιτική αυτό έχει σημασία. Ένα δεύτερο σημείο. Είναι πολύ καλό αυτό που λέτε ότι ορισμένες χώρες ε, ε, αριστεύουν. Η ε, Πολωνία, ας πούμε, με πολύ σκληρή δουλειά και με χρήματα. Ποιο είναι το μυστικό των Πολωνών. Δουλεύουν πολύ, βάζουν πολλά λεφτά εκεί. Γιατί αριστεύουν. Εγώ δεν παίρνω θέση, απλώς ρωτώ. Λοιπόν, στη σελίδα 86-87 ανοίγω και βλέπω ότι στη διοικητική ικανότητα στη συνοχή έχετε βάλει έξι σημεία, έξι φορές είναι η Ιταλία και πέντε φορές έχει πρόβλημα. Τι έγινε στην Ιταλία. Ως Επιτροπή θα κάνουμε και αποστολή αρχές του έτους εκεί, μια αντιπροσωπεία μας και θα πάμε σε μια από τις περιφέρειες που κατονομάζεται, Καλαβρία. Θα πάμε λοιπόν στην Καλαβρία και εκεί μας λέτε ότι είναι έκτακτες οι περιστάσεις, ε, πολιτική παρέμβαση ε, στη δημόσια διοίκηση, αδυναμίες ε, στους θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας αδιαφορεί, προβλήματα γενικότερα. Θα συνεχιστούν αυτά. Και ποιο είναι το συμπέρασμα, ωραία τα διαπιστώνετε. Μιλάμε για τους καλούς και μιλάμε και για αυτά που χωλένουν. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεται όμως. Αφού προσέξατε, μελετήσατε τόσο πολύ τη διοικητική ικανότητα. Υπάρχει κάποια συνέχεια, αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Η πολιτική τι κάνει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευχαριστώ. Thank you. The next Ευχαριστώ. Ο κύριο Σόιτ, την επόμενη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλή είναι η ερώτησή μου. Αναφερθήκατε στις δυσκολίες πολλές φορές οφείλεται στις δεκιμάνσεις ε, όσον αφορά το προσωπικό στις διαχειριστικές υπηρεσίες. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσωπικού που οφείλονται στο προσωπικό. Ξέρουμε ότι με τις δημοσιονομικές δυσκολίες, με την κρίση, το θέμα αυτό του προσωπικού ίσως οξυνθεί λόγω μείωσης προσωπικού αποφάσεις μπορούν να πάρουν κάποιες χώρες. Πιστεύετε ότι αυτό θα δυσκολέψει τα κράτη-μέλη και τις διαχειριστικές αρχές όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Πολλές φορές πρόκειται για τεχνικά θέματα, δύσκολα θέματα. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος που αντιμετωπίζει προβλήματα προσωπικού ε, και όσον αφορά τους αριθμούς, αλλά και όσον αφορά τις δεξιότητες αυτών που καλούνται να χειριστούν αυτά τα προγράμματα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και αυτά τα προβλήματα προσωπικού μπορεί να έχουν ε, σαν ε, συνέπειες και επιπτώσεις ε, άμεσα επί των πληρωμών, γιατί αυτό διαβάζουμε στην έκθεση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα προσωπικού να μην μειώσει την δέσμευση των κονδυλίων επιτόπου στα προγράμματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριο Τσίκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Στη μελέτη αυτή της κυρίας Χάμψα φαίνεται ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την διοικητική ικανότητα, ιδιαίτερα εκείνη που αφορά τους οργανισμούς διαχείρισης Βεβαίως υπάρχει θέμα ε, ελήψεων προσωπικού και αποχώρησης προσωπικού. Γι' αυτό ίσως το θέμα της ικανότητας ε, οδηγεί σε απόρριψη επιχειρησιακών προγραμμάτων. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δούμε τις επικρίσεις που σχετίζονται στα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε η Ιταλική περίπτωση. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι σε βάθος αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω ότι μία διοικητική ανεπάρκεια δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε απόρριψη στρατηγικών και στόχων. Θα πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε με εκείνες τις ε, δραστηριότητες που οδηγούν σε διασάφιση των στόχων. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον συντονισμό των ε, διαδικασιών και δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ τοπικών κρατικών και περιφερειακών αρχών. Αλλά ίσως αυτό αφορά μία εγωιστική προσέγγιση καθαρά. Θα πρέπει να υπάρχει μία καθολική κατανόηση αυτής της γλώσσας. Αν κάποιος προτεύει, το έχει κατανόηση αυτό, όπως είναι η περίπτωση της Πολωνίας δηλαδή ασχολούμαστε με τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μόνο θα κατανοήσουμε τις προτεραιότητες αυτές και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και πληρότητα στην ανάλυση διότι στην Ιταλία ελαχιστοποιούμε αυτά τα κριτήρια ως προς το διαδικαστικό για μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοικητικής αυτής ενίσχυσης. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ιταλίας είναι ανεπαρκές γιατί η εθνική μας κυβέρνηση δεν κατανοεί τα προγράμματα αυτά ευρωπαϊκού χαρακτήρα και θα ήθελα να σταθώ σε τρία στοιχεία. Καταρχήν το ρόλο του οργανισμού συνοχής λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά δεν λειτουργεί στην πράξη. Δεν υπάρχει προσωπικό. Και επίσης αυτή η διαλεκτική σχέση μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και περιφερειακών κυβερνήσεων δεν έχει διασαφιστεί και επίσης ε, το ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να οδηγήσει σε μια ρήξη με το παρελθόν, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει μία ε, συνέχεια σε αυτή την ε, τυποποίηση όπως ορίζεται από το σημείο 10. Δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να υποκαταστήσει αρχές που διαχειρίζονται περιφερειακά ζητήματα. Αυτό όμως δεν ισχύει και θα ήθελα να μου πει η ε, κυρία Χάμσα πόσο μπορούν να διορθωθούν αυτά τα στοιχεία ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι επικρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαλέτιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την μελέτη σας, πολύ σημαντική, με πολλά στοιχεία που απορρέουν από τις έρευνές σας. Διαβάζω ότι τα κράτη-μέλη ξεκίνησαν πολύ νωρίς την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Και εδώ λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και το αντίστοιχο έγγραφο. Έχω την εντύπωση ότι κάτι λείπει όμως από αυτήν την ε, μελέτη και από τα πορίσματά σας. Τα κράτη-μέλη σίγουρα πρέπει να έχουν διαφορετική στάση έναντι αυτής της πολιτικής συνοχής, παραδείγματος χάρη όσον αφορά την αναπτυξιακή πλευρά αυτής της πολιτικής συνοχής. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό χωρίς να περιμένουν και να έχουν κατά νου τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι τα κράτη-μέλη γνωρίζουν τις ανάγκες τους όσον αφορά την ανάπτυξη, όσον αφορά την συνοχή. Και βεβαίως υπάρχει από εκεί και πέρα, υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης και δεν είναι μόνο ε, τα κονδύλια που προέρχονται από την πολιτική συνοχής. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται λοιπόν καλύτερη επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, έτσι ώστε να εξηγήσουμε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρόλος που πρέπει να παίξουν τα κράτη-μέλη, να εκφράσουν τις ανάγκες τους που μόνο τα κράτη-μέλη γνωρίζουν και να περιμένουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σίγουρα θα έρθει αργότερα. Χρειάζεται πολιτική συνοχής σαν κάτι που δεν είναι παράλληλο με αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και έκφραση των αναγκών από μέρους των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έντεριτς. Ευχαριστώ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπατε. Μιλάτε για τις δυσκολίες, έτσι ώστε να περάσουν τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Ίσως θα ήταν πιο εύκολο να δούμε πώς ε, γίνεται αυτή η επικοινωνία και θα μπορούσε να γίνει και αμφίδρομα. Όσον αφορά τον εθνικό σχεδιασμό και προγραμματισμό και όσον αφορά, αν θέλετε, αυτόν τον σχεδιασμό και την ανεξαρτησία που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, δεν αναφέρεται πουθενά κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε βεβαίως και στις ειδικέ δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ομοσπονδιακά κράτη. Αυτό το αναφέρετε κάπου ε, στην έκθεσή σας. Όσον αφορά την χώρα μου, αν κοιτάξει κανείς αρμοδιότητες των περιφερειών, των πόλεων όπως τη συγκεκριμένη πόλη του Birmingham παραδείγματος χάνει, θα δείτε κάποιες δυσκολίες. Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μεγάλη αντίσταση προς αυτήν την ιδέα. Και αν κοιτάξετε τι συμβαίνει στην Μεγάλη Βρετανία, θα διαπιστώσετε ότι ακόμα και η ιδέα αυτού του προγραμματισμού δεν βρίσκει έφορο έδαφος. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αξιολογήσω αυτό το έγγραφο που μόλις μας παρουσιάσετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, τρεις, προς τους συντάκτες αυτού του εγγράφου. Θα ήθελα να μου πείτε αν καταρχήν έχετε κάποια συγκεκριμένη γνώμη για το εξής. Υπάρχει σαφής διαφορά αποτελεσματικότητας όταν υπάρχει μία πιο κεντροποιημένη, συγκεντρωτική αν θέλετε προσέγγιση σε σχέση με την αποκεντρωμένη προσέγγιση. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπεράσματα όσον αφορά αυτήν την διαφορετική προσέγγιση ή τα διαφορετικά αποτελέσματα εξηγούνται μόνο από τις ε, πρακτικές των διάφορων χωρών. Δεύτερον, το θέμα του προσωπικού. Υπάρχει τρόπος απλοποίησης των διαδικασιών και των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και οι οποίες τελικά μας δείχνουν ότι δεν φτάνουν μέχρι τους δικαιούχους ακριβώς επειδή υπάρχουν προβλήματα προσωπικού. Τρίτον, ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία πολύ πρόσφατα δημιουργώντας μια task force όπως πρότεινε και ο συνάδελφος από την Ιταλία εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια ομάδα εργασίας, μια task force για την δημιουργία προγραμμάτων που στοχεύουν ακριβώς τις περιφέρειες. Θεωρείτε ότι αυτή η task force θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του παρατηρητή, να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις χώρες και τις περιφέρειες που συνεχίζουν και έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξής. Προσωπικά πιστεύω ότι η μελέτη σας είναι πάρα πολύ σημαντική όσο και απαραίτητη, διότι θα πρέπει να ξέρουμε πώς ε, έχουν προετοιμαστεί τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα της νέας περίοδου 2014-2020. Πολλά σχόλια ακούσαμε, πολλές ε, προτάσεις Κατά την άποψή μου, όλα αυτά ε, και θα εισακουστούν και θα εφαρμοστούν. Μας είπατε ότι υπάρχουν χώρες, εκείνες δηλαδή που έχουν ισχυρές περιφέρειες και ισχυρές περιφερειακές δομές, ε, που είναι κράτη αποκεντρωμένα ή ομοσπονδιακά, έχουν καλύτερες επιδόσεις. μελετήσατε 7 χώρες και η Φιλανδία και η Εσθονία δεν έχουν τέτοια διάρθρωση και μάλλον δεν έχουν και περιφερειακή δομή. Θεωρούνται μία περιφέρεια, η χώρα ολόκληρη. Ποιες λοιπόν είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Αυστρία και την Εστονία. Θα με ενδιαφέρε να δω τι έχετε διαπιστώσει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια χώρα που έχει ομοσπονδιακή δομή και μια άλλη που δεν έχει καθόλου περιφέρειες προσωπικά συμμετείχα στο πρόγραμμα ε, στη Λιθουανία την περίοδο 2007-2013. Έχω ιδία πείρα και νομίζω ότι ε, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει πραγματικά να συνεργαζόμαστε ε, σε τοπικό επίπεδο και να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές ήδη από την αρχή ε, την περίοδο της διαπραγμάτευσης. Όχι να βγαίνει μια κεντρική κυβέρνηση και να βγάζει φυρμάνια και να λέει θα το εφαρμόσετε τώρα, γιατί έχετε αυτή την εντολή και αυτά τα χρήματα. Άμεση συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης, εάν κατά τη διάρκεια της μελέτης κοιτάξατε και το ρόλο των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, πάντα εξάντε, δηλαδή στο πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα 2014-2020, στο στάδιο της διαπραγμάτευσης και όχι πλέον της υλοποίησης λιμένων αποφάσεων. Μιλήσατε για προβλήματα ελλείψης και προσωπικού και επιδόσεις και πιστεύω ότι και η Λιθουανία πλήττεται από αυτή τη μάστιγα. Μιλήσετε και για χαμηλούς μισθούς. Και ε, ο κόσμος που ασχολείται με αυτά τα προγραμμάτα απασχολείται και ένα χρόνο ή δύο και μετά φεύγει. Πάει να βρει αλλού δουλειά καλύτερη. Μήπως θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα ποσό για τους μισθούς για να μπορέσει το προσωπικό να παραμένει σε αυτές τις θέσεις. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστούμε, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να μας απασχολήσουν και αυτά τα θέματα και να δούμε την κατάσταση για να τη μελετήσουμε σε όλες τις χώρες και στις 28 για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλάβουν και τα κράτη-μέλη που βρίσκονται. Αναφέρεται την Πολωνία ως καλό παράδειγμα και την Αυστρία, αλλά θα είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε μια συνολικότερη μελέτη. Κυρία Κρέλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έχασα τη μελέτη, γι' αυτό κοίταξα τώρα το κείμενο με τις διαφάνειες. Την ίδια συζήτηση είχαμε κάνει πριν από 7 χρόνια. Λυπάμαι πολύ, εγώ είμαι εδώ παλιά καραβάνα, αλλά ε, ορισμένες συζητήσεις επαναλαμβάνονται. Είναι, ε, παραμένουν οι διοικητικέ αδυναμίες, οι ασυμβατότητες ε, των περιφερειών, των κρατών μελών και των στόχων. Ολόκληρη η στρατηγική της Λισαβόνα εκεί να βάγισε. Και έτσι παρόδο να πω το εξή. Κοιτάξτε, γενικά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην λέμε τα ίδια κάθε 7 χρόνια, πανομοιότυπα. Δεν ισχύει ότι δεν θέλουν τα χρήματα οι περιφέρειες, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε στο Μπέρμιχαμ ισχύει αυτό. Αυτό είναι ε, εφεύρεση δική σας. Επινόηση. Βεβαίως και θέλουν τα χρήματα οι περιφέρειες, διότι πολλές φορές είναι ε, τα μοναδικά χρήματα για επενδύσεις στην περιφέρεια. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε ε, ε, τις περιφέρειες με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Ίσως εκ των προτέρων στην ενδιάμεση αναθεώρηση να μας απασχολήσει αυτή η ιδέα. Να μην κάνουμε αυτή την πολιτική ε, κάθε 7 χρόνια να θέλουμε να την αλλάζουμε με νέες δυνατότητες, με νέες ρυθμίσεις, με νέους κανόνες. Με αυτή τώρα την προγραμματική περίοδο κάτι ξεκινήσαμε, εταιρική σχέση. Το είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι ήδη, εταιρική σχέση. Ε, λαμβάνεται για πρώτη φορά σοβαρά υπόψη. Λέμε ε, ευθύ εξ αρχή ότι δεν θέλουμε να τα ανατρέψουμε όλα στη διοίκηση, αλλά παραμένουμε σε αυτό που έχουμε τώρα συμφωνήσει, για τους στόχους μπορούμε να τους ξαναδούμε. Είτε είναι αυτές τώρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια μπορούμε να ξαναδούμε αν εκεί πρέπει να εστιάσει και να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό ε, το δέχομαι. Μπορεί να χρειαστεί συζήτηση, αλλά μην αλλάζει συνέχεια η διοίκηση και το management, οι κανόνες γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό σας το λένε, ρωτάω, οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της μελέτης ενδιαφέρονται για να έχουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να μην ερχόμαστε κάθε 7 χρόνια να αλλάζουμε τη διοίκηση. Αυτό θα απελευθερώσει και κάποιους πόρους και κάποιες ικανότητες και θα παρακαλούσα αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμάτο. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και συμμερίζομαι τα αποτελέσματα της ε, μελέτη Σημερίζομαι ιδιαίτερα τα αποτελέσματα που αφορούν την Ιταλία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κακοδιαχείριση και όχι επαρκής διοικητική ικανότητα έμπρακτα. Και δεν ανταποκρινόμαστε στη θέληση των ε, πολιτών. Αυτό και από οικονομικής και από κοινωνικής πλευράς και ε, διαπιστώνουμε την ε, κακοδιαχείριση αυτή ως προς την ικανότητα και στον προγραμματισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να βρούμε μία νέα στρατηγική που να σχετίζεται με τα αποτελέσματα. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα καλύτερα μέσα για την εποπτεία, ιδιαίτερα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μία μελέτη σε σχέση με την ε, εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τους δημόσιους διαγωνισμούς, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ιταλία, καθώς και μία νέα μελέτη για την ανιχνευσιμότητα των, των πληρωμών για τους δείκτες σε σχέση... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βόν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, γιατί και εγώ έφτασα αργά. Έχασα την παρουσίαση και την αρχή της συζήτηση. Θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς υπογράψαμε την ε, εταιρική σχέση, συμφωνία εταιρικής σχέσης τέλος Οκτωβρίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πριν το, τέλος, πριν το τέλος του μήνα. Η περιφέρεια της Ουαλίας θα έχει ολοκληρώσει λοιπόν πριν το τέλος του μήνα το θέμα των ε, συμμετεχόντων σε αυτόν τον προγραμματισμό όσον αφορά και τη ε, χρηματοδότηση. Έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας συμπεριλαμβάνοντας 39 συγκεκριμένους οργανισμούς. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ μιας πιο συγκεντρωτικής προσέγγισης και διαχείρισης καθώς και της αποκεντρωμένης προκέγγισης. Κάποια πράγματα πρέπει να αποφασίζονται σε επίπεδο κρατών μελών και βεβαίως πολλές φορές βλέπουμε αλλαγές και δομή στο εσωτερικό των κρατών μελών. Αυτό συμβαίνει μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις δικές μας περιφέρειες ή είναι κάτι που συμβαίνει και αλλού και αυτό σίγουρα επηρεάζει την διαχείριση των ε, διαρθρωτικών πόρων, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο όνομα είναι ο κ. Μπόκοβιτς, ε, στον κατάλογο μιλτών. Σας ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά διάβασα αυτήν την ε, μελέτη, την οποία βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτά τα οποία μας παρουσιάζεται, παρουσιάζονται με εξαιρετικά ξεκαθαρό τρόπο και στη Σλοβενία. Αναφερθήκατε στην πολιτική αστάθεια στη Σλοβενία τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Εγώ ο ίδιος ε, πέρασα από πάρα πολλά διαφορετικά πόστα. Ήμουν δήμαρχος για τέσσερα χρόνια, υπουργός, ήμουν στην αντιπολίτευση και βεβαίως ε, αυτό μας δείχνει ότι το πολιτικό σκηνικό ήταν αρκετά ασταθές. Το πρόγραμμα, η προγραμματική περίοδος 2007-2013 και οι δημοσιονομικές προοπτικές σίγουρα επηρεάστηκαν και αυτό σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Νίστελ Ρόι και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν όλα αυτά τα προγράμματα μπορούμε να τα διαχειριστούμε και σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της περιφέρειας ε, και του κράτους, δηλαδή σε επίπεδο επιχειρήσεων, οργανισμών. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε διαδικασίες που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι περίπλοκες διαδικασίες. Αυτό δυσκολεύει πολύ συγκεκριμένα την ε, διαχείριση σε ένα τοπικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Στη Σλοβενία, παραδείγματο χάρη, το 2014 και το 2013, τα μέσα από την που προέρχονται από την πολιτική συνοχή ήταν πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα που οφείλονται στην κρίση και στην ύφεση. Θεωρώ όμως ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σίγουρα θα πρέπει κάτι να γίνει παραπάνω. Ο κύριος Αγημό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν εδώ ότι η πολιτική συνοχή και η διαχείριση των πόρων έχουν άμεση σχέση. Και αυτό το διαπιστώνει η μελέτη και είναι και ένα γενικό συμπέρασμα που νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουμε προβλήματα υλοποίηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση. Και στην μελέτη σας αναφερθήκατε στον έλεγχο, στους μηχανισμούς ελέγχου και λογιστικού ελέγχου που παρουσιάζουν αδυναμίες και ελλείψεις. Εγώ είμαι εισηγητής ε, της γνωμοδότησης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πολλά τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Όλες αυτές οι απάτες, οι μη κανονικές διαδικασίες που παρατηρούνται θα μπορούσαν να αποφευχούν να μειωθούν εάν υπήρχε ένας καλύτερος εκ των προτέρων εξάντε έλεγχος. Άλλη μια ερώτηση. Όλες αυτές οι παρατυπίες αυξάνονται και αυτό σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων, η αλλαγή των κανόνων από το 13 ε, με την νέα προγραμματική περίοδο βελτίωσε τα πράγματα. Μειώθηκαν αυτές οι παρατυπίες. Ή μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των αριθμών των παρατυπιών με τους νέους κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Κυρία Χάμτζα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε κάποιες από τις ερωτήσεις, αυτές που μπορείτε να απαντήσετε, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τα συμπεράσματα της ε, έκθεσής σας. Έχετε το λόγο κυρία Χάμτσα. Oh, I'm sorry. <laughs> First... Λοιπόν, καταρχάς θα απαντήσω για τη μεθοδολογία. Δεν ήταν εμπειρική αυτή η μελέτη δεν μας επέτρεπε ε, ο προϋπολογισμός να φτάσουμε μέχρι τον τελικό δικαιούχο. Παρόλα αυτά έχουμε κάνει πολλές μελέτες και ξέρουμε, έχουμε εμπειρία για την γνώμη των δικαιούχων. Και αυτό βέβαια επηρέασε και τα συμπεράσματά μας. Δεύτερον, η ιδέα ε, της μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι συστάσεις αυτές να συμπεριληφθούν σε ένα έγγραφο ε, που έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλές συστάσεις που έχουμε να κάνουμε για τα, στα κράτη-μέλη και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές που δεν χωράνε ούτε σε 100 σελίδες. Γιατί το, το βασικό πρόβλημα δεν λύνεται σε αυτό το επίπεδο, λύνεται μόνο σε επίπεδο κρατών μελών, με πολύ διαφορετικούς τρόπους και κάθε χώρα διαφέρει από την επόμενη. Αυτό για τη μέθοδο που ε, ακολουθήσαμε. Ποιο ήταν το υλικό που χρησιμοποίησαμε. Πολλές μελέτες από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής ε, Ρίτζιο, που έχουν πιο ευρύτερη εμπειρική προσέγγιση, συν επιπλέον συνεντεύξεις με τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς. Δεν ε, ρωτήσαμε όντως τελικούς δικαιούχους, αλλά έχουμε ένα δίκτυο ε, εμπειρογνωμόνων ε, που αξιολογούν, έχουν πολύ καλή γνώση της κατάστασης και τους εμπιστευόμαστε για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουν. Επίσης, ε, συνεταίρος μας, ας πούμε, είναι το EPRC, που είναι το ε, ε, αντίστοιχο Ινστιτούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση εκεί και στη βόρεια-δυτική Αγγλία, αλλά και Ευρώπη γενικότερα. Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω στα υπόλοιπα όσο μπορώ και όσο πιο δομημένα και διαρθρωμένα τα έχω σημειώσει. Για τις αλλαγές στο προσωπικό και κατά πόσο είναι κατοχυρωμένα τα διαστατικά ταμεία. Αυτό κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να το αποφασίσει μόνο του. Στην Πολωνία ε, έχουμε αυτή την ιστορία της διαρθρωτικής αλλαγής και του μετασχηματισμού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Πολωνία ήταν αναγκασμένη να αλλάξει έτσι κι αλλιώς και αυτό είναι θετικό. Έχουμε και την Αυστρία με ένα πάρα πολύ μικρό προπολογισμό σε σχέση με τον κρατικό για τα διαρθρωτικά ταμεία. Οπότε η προθυμία να αλλάξει οτιδήποτε εκεί ε, γιατί δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και να υποστηριχθεί. Τα κράτη που έχουν λιγότερα χρήματα βεβαίως το χρειάζονται και τον χρησιμοποιούν και τον απορροφούν αλλά ε, δεν θέλουν τώρα να ανατρέψουν τελείως και την εθνική νομοθεσία ε, στο βωμό των περιφερειακών προγραμμάτων. Αυτό για το κατά πόσο έχουν κατοχυρωθεί αυτά. Α, για το προσωπικό τώρα και τις αλλαγές ευθύνεται γι' αυτό ένα σύνολο παραγόντων. Βεβαίως έχουμε την οικονομική κατάσταση σήμερα που μπορεί να μην μετακινείται πάρα πολύ ο κόσμος γιατί θέλει να έχει ασφαλείς θέσεις ε, ε, εργασίας στη διοίκηση. Από την άλλη όμως οι διοικήσεις έχουν νέους κανονισμούς που κάνουν περικοπές και ε, προσλαμβάνουν μόνο για μία διετία. Σε ορισμένα κρατημέλη έτσι είναι τα νέα συμβόλαια, δεν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και οι διαχειριστικές αρχές, ας πούμε, εργοδοτούν για δύο χρόνια ένα προσωπικό και μετά χρειάζεται ανανέωση συμβολέου ή φεύγει. Ο κόσμος να πληρώνεται καλύτερα ή να έχει πιο ασφαλή θέση εργασίας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι μεταβολές στο προσωπικό. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, τον οποίο Έχω, ζητήσει, έχω ζήσει συγγνώμη, στη Βαλτική. Μια μεγάλη εταιρεία παροχής συμβουλών προσφέρει μια θέση εργασίας σε κάποιον που έχει εργαστεί προηγουμένως μετά από μια διετία, ή τριετία σε ένα διαχειριστικό φορέα. Οπότε επειδή έχει τέτοια γνώση και τέτοια εμπειρία, πάνε εκεί και τον προσλαμβάνουν και του δίνουν και δεκαπλάσια λεφτά. Δεν μπορεί ποτέ μια διαχειριστική αρχή να ανταγωνιστεί ε, μια μεγάλη τέτοια εταιρεία παροχής συμβουλών. Τώρα, για την Ιταλία, που έχει ακουστεί επανειλημμένα. Νομίζω είναι ειδική περίπτωση. Έχει πολλά επιχειρησιακά προγράμματα και οι περιφέρειες είναι πολύ ισχυρές. Εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα τα ιταλικά θέματα από μένα, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία κράτους περιφερειών. Ιδιαίτερα στην Ιταλία. Θα θέλουν βοήθεια οι περιφέρειες και πολύ ε, στενή παρακολούθηση στην εφαρμογή. Τώρα, η θεματική επικέντρωση της νέας προγραμματικής περίοδου ε, βοήθησε πάρα πολύ για να εστιαστούν τα προγράμματα και να αποφευχθούν έτσι, πώς να το πω, κατακαιρματισμένα προγράμματα σε όλες τις περιφέρειες. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναφέρθηκε τα εκάστοτε ΕΣΠΑ, ας πούμε, αναφέρουν αναλυτικά τα διάφορα προγράμματα. Και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη τώρα. Το είπα και προηγουμένως. Οι όροι που τίθενται εκ των προτέρων, οι λεγόμενοι εξάντε αιρεσιμότητα. Πολλά κράτη ε, εκφράζουν επικρίσεις βέβαια για αυτά, αλλά είναι ένα εργαλείο αυτό ένα μέσον για να υπάρχει καλύτερη ε, στρατηγική κατοχήρωση στους θεσμούς των διαρθρωτικών ταμείων, αν εφαρμόζονται με το σωστό τρόπο και αν βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι χώρες να τα εφαρμόσουν σωστά. για τις συνεντεύξεις που ζητούν να είναι τα συστήματα και αρχές σταθερά, ναι, εκφράστηκε ένα μεγάλο παράπονο. Ότι θα όλα κάθε φορά. Τρομάζουμε να προσαρμοστούμε και μετά έρχεται ένας νέος κανονισμός να ε, εκτοπίσει τον προηγούμενο. Μα στην ουσία στις διαρθωτικές αλλαγές δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ακόμα και μειώθηκαν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Εντάξει, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία συγκεκριμένα, έχει κάνει μεγάλη διορθωτική αλλαγή. Αλλά σε άλλες χώρες το, το, το σύστημα που διαχειρίζεται το διοικητικό αυτά τα θέματα παραμένει ακριβώς το ίδιο. Διαφθορά, Έχω την αίσθηση και πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αξιολογήσεις. Στην Αυστρία, ας πούμε, δεν ξέρω καμία άλλη χρηματοδότηση που να ελέγχεται ε, σε τέτοιο βαθμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ή λιγότερη διαφθορά σε άλλα προγράμματα γιατί δεν υπάρχει συστηματική αξιολόγηση σε καμία άλλη χρηματοδότηση, εθνική ή περιφερειακή. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει ε, έλεγχο και αξιολόγηση και είναι καλό αυτό ως βέλτιστη πρακτική να εφαρμόζεται και σε άλλες πηγές και σε άλλα ταμεία. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι στην Αυστρία έχουμε πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα και δεν είναι όλα διαφθορά. Πολλά σφάλματα γίνονται, λάθη κανονικά. Το ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά κάθε παρατυπία δεν είναι συνώνυμο της διαφθοράς. Υπάρχει και πρόβλημα καμιά φορά ερμηνείας ε, ανάμεσα στο δικαιούχο, στη διαχειριστική αρχή, στη δευτεροβάθμια ελεκτική αρχή. Ενέχονται εκεί πολλοί και γίνονται και παρεξηγήσεις και πολλές φορές οι εθνικές αρχές έρχονται να επιβαρύνουν με δική τους νομοθεσία ε, το πώς ε, γίνεται ο οικονομικός έλεγχος και η οικονομική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Μεγάλη αλλαγή δεν περιμένω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρξει σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. What else? Sorry. Yeah, the public procurement. Α, για τους διαγωνισμούς, τις δημόσιες προμήθειες, ναι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι... Ε, Είμαστε κάτω από το όριο της εθνικής νομοθεσίας. Υπάρχουν χώρες που έχουν ακόμα και περιφερειακή νομοθεσία που έρχεται να προσθεθεί στην εθνική και την ευρωπαϊκή για τις δημόσιες προμήθειες. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε και μέχρι 500 ευρώ προκήρυξη αγωνισμού. Αυτό και χρόνο ε, τρώει και είναι και πάρα πολύ βαριά διαδικασία. Και ενθαρρύνει τον κόσμο να παρακάμπτει τη διαδικασία. Ας πούμε, Παράδειγμα, στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, άλλαξαν τις διαδικασίες για τις δημόσιες προμήθειες για μια καλύτερη εφαρμογή στο, ε, ε, του Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης και του επιχειρησιακού προγράμματος. Για μένα αυτά είναι θέματα κρατών δηλαδή θα πρέπει οι δημόσιες συμβάσεις να ε, είναι προσαρμοσμένες στην εκάστοτε πραγματικότητα και προβληματική. Διαφέρει πάρα πολύ η κατάσταση και η προσέγγιση από χώρα σε χώρα. What else? Τίποτα άλλο. Yeah, and, I Για τις χώρες που είναι πιο αποκεντρωμένες ή πιο συγκεντρωτικές. Πρώτον, δεν μπορεί κανείς να πει ότι μια αποκεντρωμένη δομή είναι πιο δύσκολη από μια κεντρική. Η Πολωνία, ας πούμε, είναι αποκεντρωμένη. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο ως προσέγγιση. Και η Γερμανία εκ των πραγμάτων ε, έχει περιφερειακή προσέγγιση γιατί μεγάλες χώρες οδηγούνται σε αυτό μοιραία. Από την άλλη η Λετωνία και η Εστονία είναι μικρές χώρες και δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη να κάνεις και περιφερειακή πολιτική προσέγγιση. Βέβαια και η Αυστρία είναι μικρή χώρα. Στην Εστονία και παρακαλώ να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Δεν είναι πολύ ισχυρό ομοσπονδιακό το σύστημα όπως είναι στην Αυστρία. Που στην Αυστρία η ομοσπονδιακή δομή κυβερνάει τη χώρα. Δεν μπορείς να ε, συγκεντρώσεις αυτές τις προσπάθειες στην Αυστρία. Διότι είναι πολύ μικρός ο προϋπολογισμός που δεν έχει νόημα να ε, διαιρεθεί δια του 8 που είναι το ομόσπονδα ε, κρατήδια στην Αυστρία. Αυτό είναι το θέμα. Με ποια αποτελεσματικότητα, σε ποιο επίπεδο θα εφαρμόζουμε, θα εκτελούμε ένα προπολογισμό. Αυτή είναι η αντίθεση, όχι μια διαλκυστίδα περιφερειακών αρχών κεντρικών. Ε, η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα δώσω το λόγο τώρα σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Πέρεν. Ε, ο κύριος Μπόιμαν. Thank you, thank you. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μπόιμαν και είμαι αρμόδιος για την παρακολούθηση αυτής της πολιτικής. Εργάζομαι εδώ και 1,5 χρόνο στο τομέα αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για τη μελέτη σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα στα οποία φτάνετε και πάρα πολύ χρήσιμα για μας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα θέματα και πιστεύω πραγματικά ότι όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα και όσον αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες ε, έχουμε συνεργαστεί για πάρα πολλές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, αλλά τις διαδικασίες που αφορούν αυτές τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Όσον αφορά τις ε, αδυναμίες, τα προβλήματα, τα διέξοδα που διαπιστώσαμε και εντοπίσαμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Ζητήσαμε από τις ε, αρμόδιες κρατικές αρχές ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που θέλουν να υιοθετήσουν και για ποιο λόγο, τι πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί με αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δημιουργήσαμε λοιπόν τρεις Θεωρούμε ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε την διοίκηση και τη διαγύριση, πρέπει να μειωθεί ο αριθμός καταρχήν των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται η κάθε αρχή και εδώ προκύπτει βεβαίως το θέμα του προσωπικού. Υπάρχουν κράτη-μέλη, αυτά που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και αργότερα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα προσωπικού. Ο τρόπος λοιπόν πρόσληψης, κατάρτισης του προσωπικού είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον πυλώνα. Και βεβαίως συστήματα αξιολόγησης, συστήματα συντονισμού και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα και αυτά τα συστήματα αξιολόγησης για να ενισχύσουμε την διοικητική ικανότητα. Αυτοί οι τρεις πυλώνες θα πρέπει να υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο ταυτόχρονα. Αλλά βεβαίως το θέμα της διακυβέρνησης δεν καλύπτεται πλήρως από αυτές τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Πώς οργανώνεται η διακυβέρνηση, σε πολιτικό, περιφερειακό επίπεδο. Και βεβαίως εδώ το θέμα της πολιτικής αστάθειας και της διαφθοράς παίζουν ένα μείζωνα ρόλο. 27 από τις 28 συμφωνίες εταιρική σχέσης έχουν προχωρήσει και βεβαίως θέλουμε αυτές οι συμφωνίες να μεταφραστούν και να μεταφερθούν στην πράξη μέσω πολύ συγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα τεχνικά προβλήματα που μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν από τα κράτη-μέλη κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους σήμερα περνάνε από πιο ενοποιημένες και εναρμονισμένες διαδικασίες. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των τεχνικών προβλημάτων. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ερεσιμότητας, όσον αφορά τις εξαιρέσεις ε, που υποβάλλουν κάποια κράτη-μέλη και τα αδιέξοδα και τις αδυναμίες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπιστούν. Ξέρουμε ότι η τεχνική υποστήριξη υποβάλλεται κυρίως σε τομείς όπως τον τομέα του προσωπικού, της κατάρτισης, την στήριξη για περισσότερες προσλήψεις, ε, όπου εδώ βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα χρηματοδότησης των μισθών και της κατάρτισης αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα για τους πιο σημαντικούς δικαιούχους. Προτείνουμε να μας υποβάλουν ένα σχέδιο για το πόσα άτομα χρειάζονται, πόσους θέλουν να προσλάβουν και για ποιους τομείς. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε τώρα σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης της νέας γενιάς προγραμμάτων. Πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί για θέματα όπως οι κρατικές προμήθειες, παραδείγματος χάρη, τα ενδιάμεσα σώματα, οι ενδιάμεσοι οργανισμοί και φορείς, οργανώνουμε σεμινάρια σε 10 κρατημέλη με θέμα την καταπολέμηση της απάτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, μελέτη που μας παρουσιάσατε και για τα σχόλια και τη συνεισφορά της Κομισιόν. Θα Τους επόμενους μήνες θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ζητήματος για να δούμε πώς ε, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών και επιτροπής και τα αποτελέσματα, να δούμε και τα αποτελέσματα της μελέτης και της εξελίξης σε κάθε κράτος σε σχέση με, το, με τα θέματα της συζήτησής μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η ετήσια έκθεση για το 13 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταπολέμηση της απάτης. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει συντάξει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας μετά από την έκθεση του 13 της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Αριμό είναι ο συντάκτης. Η ΕΚΟΝ ζήτησε γνωμοδότηση, η δική μας γνωμοδότηση μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Ε, είναι στενό το χρονοδιάγραμμα βεβαίως και για να ε, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ε, χρειάστηκε να αποστείλουμε προσχέδιο γνωμοδότησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γι' αυτό και δεν υπήρξαν μεταφράσεις εν Γι' αυτό λάβατε το σχέδιο γνωμοδότησης στα αγγλικά. Οι μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Προτείνω λοιπόν το εξής χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες μας. Θα λάβετε το μεταφρασμένο κείμενο μέχρι τις 7 Νοεμβρίου θα αποφασίσουμε ενδεχομένως να έχουμε μία προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις 13 ε, Νοεμβρίου, ημέρα 5η δηλαδή μία εβδομάδα μεταξύ λήψης των μεταφράσεων και τελικών, ε, τελικής προθεσμίας και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στη συνάντηση της Επιτροπής μας στις 3 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η πρόταση χρονοδιαγράμματος και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρημού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η σημερινή έκθεση αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, συγκεκριμένα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή καθ' αυτή ως έγγραφο, σελίδες πολλές. Το είπατε κι εσείς, θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι η Επιτροπή Προπολογισμών θα δώσει τη δική της νομοδότηση προσεχώς. Εγώ δηλαδή ε, είχα μια εβδομάδα για να κάνω όλη αυτή τη δουλειά και είναι πολύ λίγη η προθεσμία που έχουμε για τις ε, τροπολογίες. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας παρουσιάσω την νομοδότηση που είναι σύντομη και τι προσπάθησα να πω και να εξηγήσω. Γιατί θέλω Βεβαίω και μπορεί να συμπληρωθεί και να τροποποιηθεί από την Επιτροπή. Μιλούμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και για καταπολέμηση της απάτης. Όλοι συμφωνούμε, πιστεύω, ότι θα πρέπει να είναι χρηστή η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λογικό, έτσι δεν είναι. Και όποιος έχει αυτή την προσεκτική και χρηστή διαχείριση και το λέει, αυξάνει και την αξιοπιστία ε, των ε, θεσμικών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν χειρίζεται αυτά τα χρήματα. Τώρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων ε, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ένα κράτος μέλος δεν φαίνεται πάντα πρόθυμο να δηλώνει τις παρατυπίες, ατασταλίες ακόμα και απάτες, γιατί αυτό θα έχει ε, επιπτώσεις. Είτε θα χειροτερεύουν οι στατιστικές χώρες είτε θα τους αφαιρούν ακόμα και κονδύλια. Αλλά ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την καταπολέμηση αυτών των παρατυπιών και των απατών που θα πρέπει νωρίς να εντοπίζονται και να βγάζουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Αυτό συνεισφέρει και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη φορά είναι κάπως αρνητική αυτό τον καιρό και μπορεί να βελτιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Πολύ συχνά συζητούμε για τα 23 δισεκατομμύρια που εκκρεμούν σε πληρωμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μια κακή εικόνα αυτή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα πρέπει εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια τα χρήματα που μας εμπιστεύονται ε, στα χέρια μας και στα κράτη των κρατών μελών να τα διαχειριζόμαστε σωστά. Σε καιρούς και πενιχρούς που έχουμε πολύ μικρούς σφιχτούς κρατικούς προϋπολογισμούς και περικοπές ε, από το Συμβούλιο και στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Θα πρέπει να έχουμε εκεί καλά επιχειρήματα για να λέμε ότι σωστά και χρηστά διαχειρίζεται η Ένωση τα χρήματα που τις εμπιστευόμαστε για να μπορούμε να πηγαίνουμε και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό έτσι. Όποιος ασχοληθεί λοιπόν με αυτή την έκθεση, όπως έκανα και εγώ, εγώ ξέρετε είμαι νομικός και αναρωτήθηκα για θέματα έτσι ουσίας. Πρώτον, πώς ορίζεται το οικονομικό συμφέρον της Ένωσης, πώς το ορίζει η Ένωση ίδια, πώς ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απάτη και πώς ορίζει την παρατυπία. Στην έκθεση γίνεται μια διάκριση και καλά κάνει. Από τη μια έχουμε τις απάτες και από την άλλη έχουμε τις παρατυπίες που δεν είναι απάτη εξορισμού αυτή. Αν κοιτάξετε λοιπόν το έγγραφο για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2012-363, εκεί ορίζεται η απάτη, αλλά στην εισαγωγή της έκθεσης ή της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαριθμείται ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η απάτη στα διάφορα όχι απάτη γενικώ και ορίστος, αλλά απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ποιες δυνατότητες επιβολής κυρώσεων υπάρχουν. Και θα έρθετε να διαπιστώσετε ότι στα 28 κράτη-μέλη έχουμε 28 διαφορετικές προσεγγίσεις και λύσεις και 28 ακόμα διαφορετικούς ορισμούς της απάτης. Οπότε για μένα αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της απάτης και της παρατυπίας θα πρέπει να μιλάς για το ίδιο πράγμα. Γιατί όταν διαφέρουν τόσο πολλοί ορισμοί υπάρχουν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, παρά αυτής της πανσπερμίας ας πούμε και ε, ανιομοιογένειας της παραμέτρους έχει συλλέξει στοιχεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει καταλήξει σε αυτή την έκθεση. Οι αριθμοί και τα στοιχεία είναι του 2013 και θα προσπαθήσω να συνθέσω και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία. Το 2013 συνολικά, όλα μαζί δηλαδή αν τα συνυπολογίσεις, είχαμε 16.000 παρατυπίες που ήταν απάτες ή και μη απάτες. Συνολικά 14 δις που ήταν δόλιες ε, ε, από τη μια παρατυπίες ή μη. 14 ε, δι συνολικά μπορεί να σας φαίνεται μικρός ε, αριθμός ε, γενικά σε σχέση με τον προϋπολογισμό, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 1,34 στις πληρωμές και 1,86 στα έσοδα. Τι σημαίνει αυτό. Κάνουμε μελέτες και μετρήσεις κάθε χρόνο για να συγκρίνουμε. Αν συγκρίνουμε λοιπόν την έκθεση του 13 με την έκθεση του 12 ή παρατυπίες αυξήθηκαν άκουσον άκουσον κατά 17%. Οι δηλωμένες περιπτώσεις αυξάνονται κατά 17%. Από την άλλη όμως, και αυτό είναι που μας εκπλήσει, μειώνεται το ποσό που εντάσσεται στην απάτη ή στην παρατυπία κατά 36%. Δηλαδή από τη μια συν 17, από την άλλη μείον 36%. Δηλαδή υπήρξαν περισσότερες δηλώσεις, αλλά λιγότερα ποσά. Η πολιτική συνοχής, μόνο για τη συνοχή μιλάμε τώρα εδώ, ε, είναι ο πολύ μεγάλος κορμός όταν ε, μιλάμε για παρατυπίες. Στην έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει αυτή τη διάκριση ε, ανάμεσα σε απάτη και παρατυπία. Απάτη είναι κάτι το οποίο έχει δόλο, μια διοίκηση και πρόθεση που παίρνει αυτά τα χρήματα νοθεύει τα έγγραφα 321 ε, ήταν αυτές 156 εκατομμύρια και από την άλλη είχαμε τις παρατυπίες που είναι σφάλμα δεν είναι σκεμμένο που μιλήσαμε προηγουμένως για την ικανότητα των κρατών μελών, δεν είναι πάντα πάτες. Υπάρχουν και παρατυπίες. λαθη λάθη. Ορισμένα αυτή την πολιτική ε, την εφαρμόζουν λάθος ή ανεπαρκώς όλο αυτό το σύνολο των κανόνων. Εξού και προκύπτουν σφάλματα. Και αυτές οι παρατυπίες είναι συνολικά για την πολιτική συνοχή 4.672 με συνολικό ποσό 1,2 δις ευρώ. 1,2 δις ευρώ από σφάλματα. Και αυτά πολλά λεφτά είναι και επίσης... Ε, απορίας άξιο. Σε σχέση με το 12, πάντα για την πολιτική συνοχή, ε, είχαμε αύξηση κατά 15% και στις περιπτώσεις απάτης αλλά και στις παρατυπίες. Και στις δύο περιπτώσεις όμως το ποσό μειώθηκε. Όπως και συνολικά, δηλαδή αυξάνονται οι αναφορές των περιστατικών των περιπτώσεων αλλά μειώνονται τα ποσά είναι περισσότερε παρατυπίε με λιγότερα χρήματα. Ωραία. Μπορεί κανεί τώρα να αναρωτηθεί και όλα αυτά τι σημαίνουν. Εάν υπάρχουν περισσότερε αναφορέ, σημαίνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης αποδίδουν καρπούς. Άρα το κράτος μέλος δεν διστάζει να αποκαλύψει ότι έχει εφαρμόσει κάποιες διαδικασίες οι οποίες πιάνουν τόπο και αποκαλύπτονται περισσότερα ή μήπως σημαίνει ότι τα κράτη κάνουν περισσότερα λάθη πραγματικά ε, στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Το πρώτο θα ήταν καλή είδηση, αλλά το δεύτερο ε, αρκετά κακή. Δηλαδή θα σημαίνει ότι το κράτος μέλος αντί να βελτιώνεται κάθε φορά στη διοίκηση και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιδεινώνεται κάθε φορά. Από εκεί πρέπει να λάβουμε μέτρα προφανώς. Από την έκθεση δεν δίδεται απάντηση στο ερώτημα αυτό, ούτε προκύπτει. Γι' αυτό και εγώ στην γνωμοδότησή μου παρέμεινα γενικόλογος και ανέφερα γενικές αρχές πρώτον που θα έπρεπε κανείς να κάνει όταν συζητούμε για παρατυπίες. Βλέπε σφάλματα. 4.700. Αυτά μπορούν να αποτραπούν, κατά την άποψή μου, αν ληφθούν μέτρα για την εφαρμογή, για την εκτέλεση, να βελτιωθεί. Έχω γράψει στη γνωμοδότηση ότι η εξάντε ε, αποτίμηση θα πρέπει να βελτιωθεί για να μειωθούν οι παρατυπίες και τα σφάλματα. Αν τώρα συζητούμε για απάτη, αλλάζουν τα πράγματα. Το κράτος δεν φέρει ευθύνη, πρόκειται για εγκληματίες. Προηγουμένως έγινε λόγος για διαφθορά. Στην πολιτική συνοχή δεν είναι διαφθορά. Όταν μιλούμε για απάτη είναι άλλα πράγματα, δεν είναι διαφθορά στις δόλιες ε, παρατυπίες. Πώς μπορούμε όμως να καταφέρουμε να μειωθεί και αυτή η απάτη. Να μην υπάρχει τόση εγκληματική ενέργεια εκεί για διασπάθηση ε, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εκεί προτείνω εγώ να ενταθεί και να ενισχυθεί ο εξωτερικό έλεγχο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προτάσει το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, προ τη σωστή κατεύθυνση κατά την άποψή μου και πιστεύει και το Κοινοβούλιο ότι είναι σωστά αυτά τα μέτρα. Πρώτον, κάποια σημεία συντονισμού τη Όλαφ. ΑΦΚΟ, Anti-Fraud Coordination Service. Δηλαδή να υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος μια τέτοια υπηρεσία για ε, να αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Όλαφ και τα κράτη-μέλη. Ή την Περιφερειακή Αρχή που είναι αρμόδια. Να λειτουργεί σωστά αυτή η θέση συντονισμού και να ε, διαβιβάζει και τα ορθά στοιχεία να μαθαίνουν τα κρατημέλη πώς συλλέγεις τα στοιχεία, τι αναφέρεις, πώς το αναφέρεις και πώς βελτιώνεται όλο αυτό. Δεύτερο μέτρο. Αυτό που είπα στην αρχή, να υπάρξει ένας νέος ορισμός επιτέλους της απάτης και της παρατυπίας. Γιατί μόνο όταν έχεις νέο ορισμό μπορείς να λάβεις και τα ορθά μέτρα για να, να αντιμετωπίσεις. Και υπάρχει και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2012-363 ε, που προτείνεται ενιαίος ορισμός για την ε, απάτη και για αντίστοιχες αξιόπινες πράξεις και για την καταπολέμησή τους. Στις 16 Απριλίου του 2014 το Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτό το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση και αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της απάτης αυτής καθ' αυτής. Και κάτι ακόμα που είναι ίσως το πιο επίμαχο, το Κοινοβούλιο το Μάρτι του 2014 συμφώνησε με αυτό το μέσο που είναι η ε, ε, ίδρυση μιας ευρωπαϊκής εισαγγελία. Και δεν λέω ένας εισαγγελέα που να ασχολείται με τα πάντα, αλλά που να περιορίζεται ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να οριστεί ποια μορφή θα έχει αυτή η εισαγγελία, αλλά θα ασχολείται μόνο με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, η εξωτερική έλεγχη δηλαδή, ενισχυμένη, αυτό θα βοηθούσε και θα ε, ε, μειώνονται οι αναφερόμενες ως απάτες ε, παρατυπίες. Και επίσης δεν θα υπάρχει και αυτή η σίγουρη συμφερόντων. Δηλαδή θα το δηλώσω ή όχι, θα είναι εις βάρος μου, θα μου κόψω τα λεφτά, γιατί να το δηλώσω. αυτό, και αυτό θα περιοριστεί. Αυτό τι σημαίνει. Ανταλλαγή ε, πληροφοριών ενημέρωση πιο εύκολη με την ΟΛΑΦ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στα σφάλματα και τις παρατυπίες και την απάτη και θα έχει και αποτρεπτικό απολύτως ε, χαρακτήρα και ε, δράση. Αυτά όλα τα αναφέρω λοιπόν στην γνωμοδότησή μου. Η πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου να κάνουμε τροπολογίες, διότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα αποφασίσει προσεχώς τη δική της έκθεση. Εμείς θα ψηφίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ η έκθεση επί της ουσίας του κυρίου Πυρίνσκη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι στις 8 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια το Φλεβάρι του 2015. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Γραμματεία για τη βοήθεια και τη συνεισφορά. Ήταν πάρα πολύ ε, μικρές προθεσμίες, τροχάδι. Και περιμένω τη δραστήρια και ε, ζωηρή συνεισφορά σας. Για να συμπληρώσουμε, να βελτιώσουμε αυτή τη γνωμοδότηση που πέρσι δεν ε, κατατέθηκε, αλλά φέτος κατατίθεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Όλα τα μέλη της Επιτροπής ήδη διαθέτουν το προσχέδιο έκθεση στα αγγλικά. Θα λάβετε τις μεταφράσεις μέχρι τις 7 Νοεμβρίου και θα έχουμε χρόνο για υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Έχετε το λόγο τώρα. Ο κ. Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ πολύ για την καταπολέμηση της απάτης, ε, ε, αυτό μάλλον αποτελεί συνεχή απέτηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς, ποιος είναι η χρηματοδοτική επίπτωση των ε, ε, διαφόρων παρατυπιών που ε, είναι απότοκες απάτης όπως και αυτές που δεν είναι. Όπως ξέρουμε πρόκειται για αύξηση κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τις μη απατηλές παρατυπίες, επίσης η πολιτική συνοχής μας δείχνει ότι υπάρχουν παρατυπίες που οφείλονται στους μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Μηχανή και όχι μέσω ποινικών διαδικασιών. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς παρατείνεται ο χρόνος κοινοποίησης των ε, περιπτώσεων απάτης και όπως ε, προελέχθη θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή νέα νομικά και διοικητικά μέτρα έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε ε, πολύ πιο αποφασιστικά αυτή τη μάστιγα. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ε, καταπολεμήσει την κακή χρήση και κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος και πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης έτσι ώστε ούτε ένα ευρώ της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης να μην βρεθεί σε χέρια που δεν πρέπει. Επίσης, επειδή ζητάμε μεγάλες θυσίες από τους πολίτες μέσα στα πλαίσια των περικοπών, και της ε, επισφαλούς εργασίας θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα που ονομάζεται απάτη. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των, ε, του δημοσίου χρήματος και Μιλάμε για πρόκληση και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να κινητοποιήσουμε περισσότερους ε, δημόσιους πόρους για να ε, υπάρχουν επενδύσεις και να δοθεί μια νέα δυναμική στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία τη στιγμή που παράλληλα δεν καταπολεμήσουμε τις περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών. Έτσι θα πρέπει να παρουσιάσουμε αποτελέσματα τα οποία είναι πιο ικανοποιητικά. Αν και υπάρχουν δείκτες που είναι πιο θετικοί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέντεριτς με έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την παρουσίαση αυτή και θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση καταπολέμησης της απάτης, αλλά από τις τοπικές αρχές μέχρι τις εθνικές μέχρι εδώ το Κοινοβούλιο ισχύουν παρόμοια ζητήματα. Δηλαδή μεγαλύτερη κυβέρνηση, μεγαλύτερα και τα προβλήματα και εδώ ε, έγινε λόγος για δημόσιο χρήμα, αλλά δεν πρόκειται για δημόσιο χρήμα, πρόκειται για χρήμα του των φορολογουμένων. Μιλάμε για 2,4 δις ε, παρατυπιών και φυσικά το ε, Ταμείο Συνοχής στο Ταμείο Συνοχής οφείλεται το 15% των παρατυπιών. Οι μεγαλύτερες απάτες προέρχονται από κυβερνήσεις. Ε, οι μεγαλύτερες κυβερνήσεις δεν αποτελούν μέλος της απάντησης, αλλά του προβλήματος και αυτό με ε, απασχολεί ιδιαίτερα αλλά η δημόσια εισαγγελία είναι μία ε, αρχή που θα πρέπει να οριστεί καλύτερα. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή δημόσια εισαγγελία θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο διότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Ο κύριος Λουέρ. Ευχαριστώ δύο θέματα θα ήθελα να θίξω ως προς την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπε και ο συνάδελφος. Εδώ θα αντιταχθούμε σαν μεγάλα κόμματα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την απάτη πολύ σοβαρά, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο ε, δημιουργώντας αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη στιγμή που δεν θα συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι καθόλου παραγωγικό. Αν δούμε αυτή τη διάκριση μεταξύ απάτης και παρατυπιών, αυτή η διάκριση με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι πολύ συχνά Πρόκειται για κάτι το εντελώς διαφορετικό, διότι οι παρατυπίες μπορεί να είναι σοβαρές, σε άλλες περιπτώσεις όμως ε, ε, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Και πολλές φορές οφείλονται σε αλλαγές ε, γραμμής γιατί πολλοί ε, θεωρείται ότι ε, δημιουργούν παρατυπίες ενώ αλλάζουν τα θεσμικά πλαίσια. Αυτό δημιουργεί μεγάλες ε, παρατυπίες και καθυστερήσεις και σε κυβερνητικούς και σε μη κυβερνητικούς φορείς. Μιλήσατε για τη σημασία της πρόθεσης αλλά και τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόθεση στην παρατυπία, υπάρχει διαφορά μεταξύ των σφαλμάτων, γιατί πολλές φορές πρόκειται για σφάλματα που αφορούν και τους δικαιούχους, αλλά και τον οργανισμό που χρηματοδοτεί. Και πολλές φορές δεν γίνεται καλή ή σωστή εφαρμογή μέσα στα πλαίσια των ε, δημοσίων προμηθειών ιδιαίτερα. Δηλαδή υπάρχει νομικό πλαίσιο, σωστό νομικό πλαίσιο, ε, σωστή ή σχεδόν σωστή εφαρμογή, αλλά ε, πολλές φορές υπάρχουν ε, διαφορετικά μεγέθη και θα πρέπει να γίνει σωστή διάκριση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παρατυπίες γενικά μερικές, θα πρέπει να τις δούμε σοβαρά, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουν, έχει γίνει κακή χρήση των πόρων. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τις τεχνικές ε, παρατυπίες διαφορετικά από τις ουσιαστικές παρατυπίες. Ελπίζω όμως αυτή η διάκριση να ισχύσει πιο σοβαρά μέσα στα νέα προγράμματα μέχρι το 2020 και να μιλάμε για πραγματική απάτη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή κατά πόσο μπορεί να κάνει αυτή τη διάκριση ή θα πρέπει να γίνουν σωστά συστάσεις για την αντιμετώπιση των απατών, αλλά παράλληλα να δούμε τους, τις παρατυπίες που δημιουργούν απλώς μικροκαθυστερήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλέκ. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να χαιρετίζω τις επιπλέον προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης που είναι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο από μέρους της Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ε, ακαιρεότητα της ε, οικονομικής μας πολιτικής και τα στοιχεία που μας παρουσιάζεται εδώ δείχνουν ότι οι περιπτώσεις απάτης ή παρατυπιών αυξήθηκαν, το συνολικό ποσό όμως που αφορά αυτές τις απάτες μειώθηκε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ενισχύθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου, κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και βεβαίως η ενίσχυση των μηχανισμών και των υπηρεσιών που έχουν σαν σκοπό την καταπολέμηση της απάτης είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε θα πρέπει να γίνει σαφής ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών των υπηρεσιών που έχουν σαν σκοπό την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Πρέπει να ξαναδούμε επίσης την σύσταση νέων φορέων όπως προτείνουν κάποια κράτη-μέλη. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες και να στηρίξουμε την αποτελεσματικότητά τους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγήτη. Πάρα πολύ καλή η παρουσίασή του, η έκθεσή του. Υπογραμμίσατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο έλεγχος εξάντε και οι αξιολογήσεις για τη μείωση των παρατυπιών. Είπατε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μία ε, ενιαία, για έναν ενιαίο ορισμό. Και αυτός ο ενιαίος ορισμός δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται με τελείως διαφορετικό τρόπο ε, ανάλογα με το που βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της πρόληψης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τις παρατυπίες. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ο τελικός δικιούχος όντως ακολουθούσε μια παράτυπη διαδικασία χωρίς όμως να το γνωρίζει. εν αγνία του. Ο τελικός δικαιούχος, έλεγε ο κανονισμός, θα έπρεπε να αγοράσει ξύλινα παράθυρα και πόρτες, ένα παράδειγμα δίνω, και τελικά κατάφερε να αγοράσει φθηνότερα παράθυρα και πόρτες από αλουμίνιο. Πολύ καλύτερα όμως όταν ήρθαν τελικά οι επιθεωρητές, θεώρησαν ότι πρόκειται για παρατυπία, καθότι ο κανονισμός ε, αναφερόταν σε ξύλινα παράθυρα και πόρτες, Παρόλο λοιπόν που το ποσό ήταν χαμηλότερο και η ποιότητα καλύτερη, επρόκειτο για παρατυπία. Ο τελικός δικαιούχος ουσιαστικά, βλέποντας αυτά τα παραδείγματα, χάνει την εμπιστοσύνη του στο ευρωπαϊκό σύστημα. Χρειάζονται λοιπόν καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη ενημέρωση για να μειωθούν τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Κύριε Ζέλλας, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Αριμών για αυτήν την εξαιρετική του εργασία. Έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε για τους ορισμούς, την απάτη, την επαρατυπία. Διαπιστώνουμε όμως ότι παρατυπίες είναι οτιδήποτε δεν ακολουθεί τον κανονισμό, τους κανόνες. Από την άλλη όμως έχουμε σφάλματα, έχουμε διαφθοριά και έχουμε και απάτες. Πρόκειται για τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο οι παρατυπίες, οι οποίες πολλές φορές, αν θέλετε, οφείλονται σε σφάλματα ή σε μη προσεκτική παρακολούθηση και τήρηση κάποιων κανόνες, κανόνων. Πρόκειται λοιπόν για κάτι τελείως διαφορετικό και όταν ε, λάβει κανείς υπόψη του την έλλειψη προσωπικού, την ασάφεια ε, κάποιων κανόνων, την αλλαγή, την πολύ συνήθεια αλλαγή προσωπικού που ασχολείται με αυτά τα προγράμματα, διαπιστώνει ότι αυτές οι παρατυπίες και τα σφάλματα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μειωθεί. Ξέρετε ότι ο τομέας της γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξης της υπαίθρου παρουσιάζει πολλές τέτοιες ε, περιπτώσεις σφαλμάτων παρατυπιών μη συμμόρφωσης με τους κανόνες, η παράληψη συμμόρφωσης και ο κύριος Αριμό παρουσιάζει πολύ σωστά αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρώ ότι Αυτό που τις περισσότερες φορές διαβάζουμε στον τύπο είναι αν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής χρησιμοποιούνται για ορθούς σκοπούς ε, στα αρμόδι, στους αρμόδιους τομείς. Παραδείγματος χάρη, είναι ένα κράτος μέλος χρηματοδοτεί την ε, κατασκευή ενός αεροδρομίου με κονδύλια που προέρχονται από την πολιτική συνοχή, από τα ταμεία συνοχή. Το θέμα λοιπόν της ορθής χρήσης των κονδυλίων στον σωστό τομέα είναι κάτι που διαβάζουμε πολλές φορές στο τύπο και που θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Εμείς εδώ ακούγοντας προσεκτικά τις προτάσεις του κυρίου Αριμών όσον αφορά τους ελέγχους από ανεξάρτητους φορείς, ε, εκ των προτέρων και ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις περιπτώσεις που ε, έχουν αναφερθεί. Για τα θέματα της διαφθοράς. Εδώ αυτό είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Τα σφάλματα όμως και οι παρατυπίες που είναι η μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων που μας απασχολούν είναι κάτι που πολλές φορές οφείλεται και στο προσωπικό. Ε, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία δεν έχει την κατάλληλη κατάρτιση, δεν γνωρίζει. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι, και αυτό είναι και θέμα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές ε, στα πλαίσια της επιτροπολογίας, το θέμα της απλοποίησης. Απλοποίηση δεν είναι μείωση των κανόνων, είναι διαδικασίες οι οποίες να είναι πιο ευανάγνωστες και να ε, στο σωστό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος βανίστελ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά για αλλαγή. Εκτός από το κείμενο ε, είναι ίσως σκόπιμο να πούμε από πού ερχόμαστε. Και στην προηγούμενη περίοδο για το ίδιο θέμα είχαμε εισηγητέ τον κύριο Τόμας Ντόιτς, τον κύριο Όλμπριχτ και άλλους, ε, που μας είπανε ότι ε, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, προγράμματα δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει υλοποιήσει, εμείς τα είχαμε προτείνει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα και τα σφάλματα και τις παρατυπίες και την απάτη. Είναι πολύ ε, προσεκτική η μελέτη. Και όσο πιο προσεκτικά κοιτάς, αν πηγαίνεις με ένα μεγεθυντικό φακό ας πούμε, ανακαλύπτεις περισσότερα. Και αυτό το κάνω και εμείς στο σπίτι με τα παιδιά μου. Όταν θέλουμε κάτι να λύσουμε το συζητάμε σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, έχουμε κάνει βήματα λοιπόν σε προηγούμενες ε, δράσεις και προγράμματα και κανονισμούς και τώρα αυτό αποδίδει καρπούς. Μπορεί να είναι λιγότερο το ποσό, αλλά είναι περισσότερες οι αναφορές και περισσότερες οι λεπτομέρειες. Γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει και απάτες και τέτοιες παρατυπίες. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση με το νέο κανονισμό. Στο σημερινό κανονισμό έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και πάλι που επιτρέπουν εγκαίρως και με καλύτερη ποιότητα να ε, έχουμε στους ελέγχους. Καλύτερη ποιότητα. Ας πούμε. Αυτό που είπε ο κύριος Τσέλερ ε, για μια γέφυρα, δεν ξέρω πώς τη λένε. Ωραία να φτιακάνει μια γέφυρα, άμα δεν περνάει αυτοκίνητο, είναι μια τρύπα στο νερό και τζάμπα λεφτά πεταμένα. Δηλαδή, στο ε, τωρινό προγραμματισμό υπάρχουν τα ε, επιχειρησιακά προγράμματα, ε, υπάρχει η εταιρική σχέση, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη γνώση, καινοτομία και τώρα όλα αυτά θα πρέπει να πάνε σε αηφόρα προγράμματα, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει και πολύ καλύτερη καθοδήγηση. Αυτό θέλω να το δω και στην έκθεση. Για να πούμε ότι αλλάξαμε τα πράγματα και τώρα έχουν αποδώσει 7. Λοιπόν, μετά από 2-3 χρόνια θα έχουμε και πάλι νέες ε, πιο λεπτομερείς αναφορές, ακόμα περισσότερο, για τις διάφορες ε, συμφωνίες για τις επιδόσεις ας πούμε μείωση στο διοξίδιο του άνθρακα κτλ. Και αν δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτά αρχίζουν οι περικοπέ. Δηλαδή είναι σοβαρά τώρα αυτά που γίνονται, έχουν σφίξει τα πράγματα. Και τέλος, στο ΣΕ, το ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα επίμαχο. Το είπε και ο εισηγητή για το θέμα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Κοινοβούλιο έχει πει τη γνώμη του ότι το θέλει. Αλλά θα πρέπει να έρθουμε να διαπιστώσουμε ότι όταν έχουμε μέσα, σαν αυτά που διαθέτουμε σήμερα, αν τα εφαρμόσουμε καλά, διερωτώμε αν χρειάζεται οπωσδήποτε και άλλο νέο θεσμό από πάνω για να κάνει την ίδια δουλειά ο εισαγγελέα. Πού είναι η προστιθέμενη αξία, δεν εφευρίσκουμε τίποτα. Απλώ εντάξει μπορεί να καταδικάζονται πιο εύκολα οι απαταιώνε, αλλά υπάρχουν και άλλα ε, μέσα. Η δήλωση αξιοπιστία, ας πούμε, που κάνουν τα κράτη-μέλη και στην συνδιαχείριση, με συγχρηματοδότηση. Υπάρχουν άλλα μέσα στη διάθεσή μας. Και ο Υπουργό Οικονομικών των κρατών μελών, του κάθε κράτους μέλους, διαπιστώνει και υπογράφει ότι είναι χρηστή η διαχείριση και βάζει και την υπογραφή του. Αυτό τι σχέση έχει τώρα με την κουλτούρα και με την νεοτροπία. Μπορεί κάποιος να έχει πιο χαλαρή νοοτροπία και να περνάνε ε, διάφορες ε, παρατυπίες και σφάλματα. Η νέα Επίτροπος Κρέτσου είπε μηδενική συνοχή. Μηδενική συνοχή. Ε, ανοχή, συγγνώμη. Αλλά πώς θα γίνει τώρα αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με ένα Ευρωπαίο εισαγγελέα για την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό που μπορούν να ρυθμίζονται στη συνδιαχείριση, στη συγχρηματοδότηση από το κράτος, από την περιφέρεια, μαζί με τη διαχειριστική αρχή, ε, μαζί με τον εκάστοτε αρμόδιο. Αυτό που χρειάζεται είναι λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτά που ισχύουν και όχι έναν απομηχανή θεό εισαγγελέα που ως διαμαγεία θα λύνει τα θέματα. Και δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Άρα καλούμε το Συμβούλιο να υποστηρίξει, λέει εδώ. Και άρα ξέρω ότι κατά πλειοψηφία δεν το θέλει το Συμβούλιο. Λέμε να υποστηρίξει το Συμβούλιο λοιπόν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν ξέρω. Πώς θα το διατυπώσουμε. Το κοινοβούλιο έχει πει τη γνώμη του, εγώ είμαι λίγο διχασμένος σε αυτό. Έχουμε λίγο καιρό να σκεφτούμε το κείμενο, θα το κάνουμε και θα κάνουμε Σε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βανίστερο. Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, quelques... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του εισηγητού, ιδιαίτερα σε ό,τι αναφέρει για το παρασκήνιο αυτής της απάτης, αλλά και για τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα κονδύλια, τους ίδιους πόρους και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Όσον αφορά την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την ιδέα για την σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελίας. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα είδαμε αμέσως ότι κάποια κράτη-μέλη και εθνικά κοινοβούλια έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες. Επίσης αναφερθείτε και ο εισηγητής στο θέμα του ορισμού της απάτης, αν είναι εσκεμμένη ε, αδικοπραγία, αν πρόκειται για παρατυπία, αν πρόκειται για οργανωμένη απάτη, δόλια παρατυπία κτλ. Όλη αυτή λοιπόν η προσπάθεια ορισμού του ε, όρου απάτης κατά τον κύριο αριμόν θα μας βοηθήσει να έχουμε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Νομίζω ότι ο ορισμός του τι είναι απάτη, πώς νοείται η απάτη, είναι κάτι που σίγουρα θα συνεισφέρει στην καλύτερη καταπολέμησή της. Ξέρω ότι ο εντοπισμός, η αναφορά της απάτης γίνεται βάσει διαφορετικών κριτηρίων από τη μία ή την άλλη χώρα και καλό θα ήταν να δούμε ποια είναι αυτά τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται ο εντοπισμός. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πιτσέρνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, πρόταση γνωμοδότησης που με βρίσκει σύμφωνη. Θα προσπαθήσω να συνεισφέρω και εγώ με ορισμένες τροπολογίες. Όπως ε, προελέχθη, η έκθεση της Επιτροπής μας δίνει μία θετική πλαισίωση της κατάστασης σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης στην πολιτική συνοχής. Έχουν αυξηθεί οι παρατυπίες, αλλά τα ποσά μειώνονται σημαντικά. Και αυτό που έχει σημασία είναι η συνεχής προσπάθεια της Επιτροπής, τους ελέγχους και στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές για την πρόληψη, όπως προελέχθη, αλλά απομένει πολύ μεγάλη εργασία επί του θέματος. Γιατί τα στατιστικά στοιχεία που μας απασχόλησαν βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια αναχώρα και είναι κατά προσέγγιση στοιχεία διότι τα στοιχεία που αποστέλλονται από τα κράτη-μέλη είναι απότοκα μίας πολιτικής πρόληψης που διαφέρει μεταξύ τους, άρα δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μία πιο λεπτομερής ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Η Ιταλία έχει επιτελέσει πολύ σημαντική εργασία που έχει τύχει εκτίμησης από την Όλαφ θα πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων λοιπόν έτσι ώστε η καταπολέμηση απάτης να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ένα ευρώ των κοινοτικών πόρων μέσα στα πλαίσια ε, ενδεχομένων απατών, ιδιαίτερα εν ώψη της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να υπάρχει καταστολή πλήρης καταστολή των απατών και γι' αυτό και οι προτάσεις Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η καταπολέμηση των απατών μέσω ποινικού δικαίου θα πρέπει να υποστηριχθούν. Ξέρω ότι κατά την προηγούμενη θητεία επιτελέστηκε μια πολύ σημαντική εργασία και στους δύο τομείς και ελπίζω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να φέρουμε το όλο θέμα σε αίσιο πέρας. Ένα τελευταίο θέμα για τις παρατυπίες που δεν αποτελούν απάτη. Ενδεχομένως θα μειωθούν εάν καταβληθεί προσπάθεια από τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια της κατάρτισης των δημόσιων αρχών για τη σωστή διαχείριση έτσι ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες στενοπούς και για να υπάρχει σωστή διαχείριση. Και εδώ μας περιμένει πολύ σοβαρή εργασία. Thank you. Thank you very... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπριό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το πολύ ενδιαφέρον έγγραφο που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, έχει πραγματικά ε, χάσει κάθε αξιοπιστία. Πώς μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν 23 δις τιμολογίων πρέπει να καταβληθούν, να πληρωθούν. Πώς μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν το 2013 16.000 παρατυπίες διαπιστώθηκαν για ένα συνολικό ποσό 2,4 δις ευρώ. Βεβαίως αυτό σχετίζεται εν μέρη με την απάτη και τη διαφθορά. Και βεβαίως ζητούμε από τους πολίτες να σφίξουν τη ζώνη και πολλοί πρέπει να υποστούν τη λιτότητα. Στη δική μου περιφέρεια, στο βορρά, στο Νόρ Παντκαλέ, βλέπουμε ότι έχουμε ανεργία της τάξης του 20-25% και δεν χορηγούνται ε, δάνεια. Δεν γίνεται όμως επαρκής έλεγχος των ε, κονδυλίων αυτών, γιατί η Επιτροπή είναι ανίκανη. Ένας ομιλητής είπε ότι στην προηγούμενη θητεία οι ίδιες προτάσεις, τα ίδια γεγονότα είχαν καταγγελθεί, αλλά τίποτα δεν έγινε για να αποφευχθεί η απάτη και η διαφθορά. Δεν πιστεύω στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι θα ήταν προσβολή προς τους λαούς και την εθνική κυριαρχία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανασταλούν οι πληρωμές και οι επιδοτήσεις στα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να τηρήσουν και να κάνουν καλή χρήση του, του δημοσίου χρήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την Επιτροπή Προπολογισμού, η οποία στην οποία συμμετέχω και στην οποία προσπαθούμε να δούμε πώς δαπανώνται και αν δαπανώνται σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως ξέρετε, με την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αυτή την εβδομάδα θα ξαναρχίσει πάλι η ίδια διαδικασία και σίγουρα θα μας αφορά και εμάς και όχι μόνο την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ σφάλματος και απάτης. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε, απάτη, σε σφάλματα ενώ ε, ουσιαστικά το ποσό των απατών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 0,2 δις συγγνώμη, 0,2% του ευρωπαϊκού προβλησμού, που είναι ένα τεράστιο βεβαίως ποσό, δεν συμπεριλαμβάνει τις παρατυπίες και τα ασφάλματα. Πρέπει να δούμε τις προβλέψεις. Πρέπει να δούμε ότι, όπως είπε πολύ σωστά ο εισηγητής, θα πρέπει εδώ να αυξηθεί, να ενισχυθεί ο ρόλος των κρατών μελών. Όπως ξέρετε υπάρχει διαφορετικό σύστημα και για την αναφορά των παρατυπιών και απατών υπάρχει διαφορετικό σύστημα διερεύνησης και εντοπισμού αυτών των παρατυπιών και των απατών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να στηρίξουμε τα κρατη εκεί όπου συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Κάθε χρόνο 4-5 κράτη-μέλη έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά ε, σφαλμάτων και παρατυπιών. Πρέπει να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε και για αυτά τα σφάλματα και τις παρατυπίες, αλλά και για τις περιπτώσεις απατών. Στηρίζω τις ε, συστάσεις του εισηγητή και θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να προσθέσω στα συμπεράσματα του εισηγητή. Η υπεύθυνα για την δαπάνη και τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι τα κράτη-μέλη. Άρα πραγματικά αυτούς πρέπει να στηρίξουμε, ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που παρουσιάζουν αδυναμίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω, σε σχέση με αυτό που μόλις είπε ο κύριος Βόγκαν, η απάτη, το πρόβλημα της απάτης, σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τους υπάρχοντες μηχανισμούς και όχι να δημιουργήσουμε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα ο οποίος ουσιαστικά προκάλεσε μεγάλες επιφυλάξεις και ανησυχίες από πολλούς όπως είπε ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετή αξιοπιστία διότι κάποιοι οδηγούνται σε απάτες. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα καταπολεμήσουμε τις απάτες. Η νέα Επίτροπος είπε ότι τα προγράμματα θα διακόπτονται άμεσα μόλις διαπιστωθεί απάτη. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή η νέα στάση της Επιτροπής θα είναι πιο αποτελεσματική. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό δημιουργώντας νέους θεσμούς όπως τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε γραφειοκρατία και πολλά έντυπα. Εάν θεσπίσουμε νέους φορείς και θεσμούς. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να αυξηθεί η αυστηρότητα των ελέγχων και η συχνότητά τους. Επίσης, να παρακολουθούμε το σύνολο των προγραμμάτων. Έχω την εντύπωση ότι τα σφάλματα που γίνονται, γίνονται πολλές φορές εν αγνία αυτών που τα διαπράττουν. Πολλές φορές επίσης λείπουν ε, καταρτισμένοι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στα νέα κράτη-μέλη, τα οποία μόλις προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία δεν έχουν ακόμα ε, σωστή κατάρτιση, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Χρειάζεται λοιπόν τεχνογνωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Α, η κυρία Μπρέσο. Ε, Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάτι σε σχέση με αυτά που προελέχθησαν. γιατί τα πράγματα διαφέρουν όταν πρόκειται για παρατυπία με βόλο, με απάτη ή παρατυπίες οι οποίες δεν οφείλονται σε απάτη και σχετίζονται με τους περίπλοκους κανόνες. Εμείς φέρουμε μεγάλη ευθύνη στον τομέα της ε, νομοθετικής απλούστευσης αλλά και στο θέμα της απλούστευσης της διαχείρισης έτσι ώστε να διαχωρίσουμε καλύτερα τις παρατυπίες ε, με δόλο, με στόχο την απάτη ή αν πρόκειται σε καθαρά γραφειοκρατικές ε, διαδικασίες του κράτους, διότι πολλές φορές τα κράτη όταν μεταφέρουν ή διαχειρίζονται την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, δυστυχώς προσθέτουν ε, και ε, άλλες περιπλοκότητες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά ακριβώς που είπε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς, για να νομοθετήσουμε καλύτερα ως προς την απλούστευση και την αρχή της επικουρικότητας, διότι πολλές φορές χρησιμοποιώντας την αρχή της επικουρικότητας απλουστεύουμε γενικότερα την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο την επόμενη θητεία να περιπλέξουμε τα πράγματα γιατί τα κράτη και ιδιαίτερα οι περιφέρειες καθώς και οι δικαιούχοι θα πρέπει να εγγυηθούν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή να καταστήσουν σαφές το τελικό αποτέλεσμα με βάση την επιμέρους ε, χρηματοδότηση και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στη γραφειοκρατία και στις διοικητικές ε, δυσχέρειες. Θα πρέπει παράλληλα με το αποτέλεσμα να απλουστεύσουμε και το διοικητικό άχθος. Έτσι θα μειωθούν και οι παρατυπίες και θα φανούν καλύτερα οι απάτες, θα φανεί καλύτερα η απάτη. Γιατί η απάτη βασίζεται σε αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να δούμε πού έγκυται πραγματικά η απάτη και με βάση τα ε, οικονομικά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τις παρατυπίες με ή χωρίς απάτη, έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα κατά πόσο πρόκειται για τεχνική παρατυπία ή πρόκειται για παρατυπία με δόλο καθαρά. Ευχαριστώ. Τώρα όμως δεν έχουμε άλλον ομιλητή. Α, έχουμε την κυρία Άντερσον. Παρακαλώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον βουλευτή που κατάφερε μέσα σε μία εβδομάδα να γράψει γνωμοδότηση για αυτό το θέμα και πραγματικά υπάρχει ένας ηρμός ε, μεταξύ των δύο τοποθήσεων και παρουσιάσεων που ακούσαμε σήμερα. Από τη μια είδαμε πώς εφαρμόζεται η πολιτική συνοχή και τα προγράμματα και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει και αυτό δεν μπορείτε να το αποσυνδέσεται από την προσπάθεια προστασίας των οικονομικών συμφερόντων. Ακούσαμε στην προηγούμενη μελέτη ότι υπάρχει πρόβλημα σε ανθρωπίνους πόρους, είναι περιορισμένοι και ε, υπάρχουν περικοπές και στους προϋπολογισμούς και στις περιφέρειες για την τεχνική υποστήριξη, οπότε δεν είναι απορίας άξιο ότι έχουμε τέτοιες παρατυπίες και κάποιες από τις πρακτικές, ορισμένες από τις περιφέρειες, χρειάζονται έλεγχο τι μπορεί να κατηγορηποιηθεί και να ταξινομηθεί ως παρατυπία. Ας πούμε, στο βορρά της Ιρλανδίας γνωρίζω ε, πολλές ομάδες που ήρθαν στο κόμμα μας και σε άλλους και ε, διαμαρτύρονται για τον τρόπο ε, που παρουσιάζονται κάποια πράγματα ως παρατυπίες. Ο καθένας θα έχει παραδείγματα. Σε μία συνεδρίαση ήρθαν 12 άτομα και ήταν πρωινή συνεδρίαση και είχαμε προβλέψει πρωινό με τσάι και ε, κουλουράκια γιατί από τους 12 να έρθουν 12 ήρθαν 11 και έγινε ολόκληρη αλληλογραφία για να δούμε ποιος έφαγε το, το δέκατο κουλουράκι ας πούμε γιατί περίσεψαν τα γλυκά αυτό είναι γελίο μπορεί να σας φαίνεται αλλά ε, μπορούν και άλλοι να σας πούνε και ότι πολλές ομάδες και οργανώσεις ε, δεν υποβάλλουν ε, ε, ακριβώς αιτήσει, γιατί μπορεί αυτό να ταξινομηθεί ως παρατυπία. Οπότε σου λέει όλες που να πάω να μπλέξω. Ακούσαμε προηγουμένως για τους περιορισμένους πόρους και οικονομικούς και ανθρωπίνους και προσπαθούμε να προσπαθήσουμε τώρα να προστατεύσουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνει όμως πραγματικά ο κατάλογος των ομιλητών. Θέλω να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εκπροσώπους της Όλαφ. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ. Ανδρέα Μπορτόνη. Είμαι από τους συντάκτες της Επιτροπής ε, για την Προστασία των ε, Συμφερόντων της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να ε, σας πω ότι εκτιμώ πολύ την ανάλυση του κυρίου Αριμών, του αξιωτήμου βουλευτού, γιατί πραγματικά βρήκε την καρδιά του προβλήματος, την κεντρική ουσία. Δηλαδή. Έχει προηγηθεί μια ολόκληρη εξέλιξη ε, τα περισμένα χρόνια και με την έκθεσή μας το 2013 προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία γιατί ήταν η τελευταία έκθεση της απερχόμενης ας πούμε Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξει μια συνολική επισκόπηση και αναδρομικά ε, να δούμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη πενταετία, κατά τη διάρκεια της θητείας της. Λοιπόν, Ακριβώς, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική προσέγγιση. Εκεί είναι ακριβώς το αγκάθι και η κυριότερη πηγή ανησυχίας. Και ο, ο ακριβής λόγος γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλά γενικά συμπεράσματα, πολύ λίγα γενικά συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και προσπαθήσαμε να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερο. Τι σημαίνει λοιπόν η διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικά νομικά συστήματα, διαφορετικά διοικητικά συστήματα και βασικούς ορισμούς νομικούς διαφορετικούς, αλλά και διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα για τα θέματα της ε, απάτης και της παρατυπίας. Υπάρχουν και διαφορετικές διοικητικές ικανότητες και στην πρόληψη, ας πούμε εδώ παρατυπιών. Επίσης, διαφορετικές προσεγγίσεις ως το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι για την ανταπολέμηση της απάτης. Και ένα τελευταίο, χωρίς αυτό να είναι λιγότερο σημαντικό, θέλω να τονίσω ότι αυτές οι διαφορές καμιά φορά υπάρχουν και στο ιστορικό του ίδιου κράτους μέλους. Ε, σε διαφορετικές διοικήσεις και μηχανισμούς του ίδιου του κράτους. Παράδειγμα, γιατί σε ορισμένες χώρες έχουμε ένα επίπεδο ανείχνευσης ε, στη γεωργία και τίποτα στη συνοχή ή το αντίστροφο. Το δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει από την πρόταση και την ανάλυση του κυρίου Αριμό είναι Πώς ερμηνεύουμε αυτή την ανείχνευση. Είναι καλή είδηση ή κακή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στην έκθεση πήραμε μια σαφή απόφαση. Από τη δική μας σκοπιά είναι καλό να ανοιχνεύονται, να εμφανίζονται αυτά τα πράγματα, γιατί σημαίνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται εξετάζονται και ενδεχομένως διορθώνονται αντιλαμβάνονται οι διοικήσει το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται και μαθαίνει το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει λύσει για να διορθωθεί. Γι' αυτό επίσης υπάρχει μια σαφής απόφαση και ένδειξη για την καταπολέμηση της απάτης. Δεν πιστεύουμε εμείς τη μηδενική ανείχνευση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το Neverland, η χώρα του ποτέ δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει μηδέν απάτες. Μηδέν απάτες δεν είναι καλό σημάδι για μας, σημαίνει ότι δεν τις βρίσκουν. Δηλαδή χώρες που έχουν αναφέρει μηδέν απάτη επί σειρά ετών, κατά την άποψή μας αποδεικνύουν ορισμένες δυσκολίες στην καταπολέμηση της απάτης. Τουλάχιστον στην ανείχνευση να τη βρούνε, να την εντοπίσουν. ή αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω, την βρίσκουν αλλά δεν την αναφέρουν. Δηλαδή κάτι πάει στραβά ακόμα σε αυτή τη ροή πληροφορία. Γι' αυτό το λόγο και με αυτόν τον τρόπο, και έτσι απαντώ εδώ στον κύριο που ρώτησε, στον κύριο Ζουλού. Έτσι, καταλήγουμε σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη με αυτή τη μεθοδολογία. Για τον εντοπισμό λοιπόν και την ανείχνευση, συμφωνώ ότι στην μεγάλη κατηγορία των παρατυπιών ε, πρέπει να γίνει διάκριση. Για παράδειγμα, ε, γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη πηγή παρατυπιών είναι η παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. Δηλαδή, αν συνδέσουμε τα αναλυτικά ευρήματα της έκθεσης με την πολιτική και την δράση, που επίσης ε, περιγράφει η έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς βασιζόμενη σε αυτές τις ενδείξεις, σε αυτά τα ευρήματα ας πούμε, έχει αναλάβει δράση και προτείνει νέες οδηγίες ας πούμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι συνομοθέτες ε, τα ανέλαβαν αυτά και το, πέρυσι βγήκε το νέο πακέτο για τις δημόσιες συμβάσεις, τις νέες οδηγίες και τώρα εναπόκειται στα κράτη-μέλη να τις εφαρμόσουν. Αυτό δείχνει πως τα ευρήματα της έκθεσης πάνε χέρι-χέρι με ε, τις πολιτικές μας και τις δράσεις. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο και πάλι κάπως λίγο κλείνω. Ε, οι πολιτικές που, που περιγράφει η έκθεση, ας πούμε ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή για την Οδηγία για την Προστασία των συμφερόντων των Οικονομικών της Ένωσης για του ποινικού δικαίου, έρχονται να απαντήσουν σε αυτές τις βασικές ανησυχίες που εξέφρασα στις αποκλήσεις, στις προσεγγίσεις διαφορετικές, ερμηνείες διαφορετική βασική ορισμή στα κράτη-μέλη για τις έννοιες ή ακόμα και διαφορετική αίσθηση και προσέγγιση για κουλτούρα απέναντι στην απάτη. Ίσως μπορώ να το πω εδώ. Είπαμε, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μηδενική απάτη. Όπου αναφέρεται απάτη μηδέν, σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη προτιμούν από την αρχή να εξασφαλίσουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά δεν καταπολεμούν την απάτη. Γιατί αν δεν επιβάλλεται κύρωση ε, στον ε, δράστη, θα βρει άλλη μέθοδο ε, και πάλι θα εκμεταλλευτεί το σύστημα και θα καταχραστεί. Δηλαδή πότε δεν πρόκειται το σύστημα να αυτοϊαθεί. Μόνο νέα προβλήματα θα παράγει και θα δίνει την αίσθηση ότι Κατά δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώ επιστρέφουμε κάποια λεπτά, λεπτά αν αυτό ανοιχνευθεί. Και ένα τελευταίο για το θέμα των παρατυπιών. Γιατί αυτό ακούστηκε πολλέ φορέ εδώ και χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνηση. Βεβαίω, είναι δύο οι πηγές των προβλημάτων. Το ένα είναι η παραβίαση των κανόνων για τι δημόσιε συμβάσει, που συνδέεται κυρίω με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν οι διοικήσεις ε, του κανόνε. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, ε, πηγή προβλημάτων είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Δηλαδή, ποια είναι η κλασική ε, παρατύπια. Κάποιες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες. Δόθηκαν και παραδείγματα. Ιδιαίτερα. Ε, κάτι με κάποιες πόρτες ξύλινες και άλλα υλικά αυτό έχει να κάνει με τη χρηστή διοικητική πρακτική περισσότερο και λιγότερο με κανόνες. Δηλαδή, αν υπογράψω εγώ με μια εταιρεία μια σύμβαση, να μου παραδώσει ξύλινες πόρτες για το σπίτι μου και επιστρέφω και βλέπω μεταλλικές, υπάρχει πρόβλημα. Ε, δηλαδή υπάρχει συμβατική υποχρέωση η οποία δεν έχει γίνει σεβαστή. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει η εταιρεία, να έρθει σε μένα και να μου πει που είμαι η δημόσια διοίκηση, που δίνω τα χρήματα, θα μου πει, συμφωνείς να μην σου βάλω ξύλινες πόρτες, να αλλάξουμε την, τους όρους της σύμβασης γιατί με βολεύει να σου βάλω μεταλλικές. Ε, όταν αυτό το διαπιστώνει κανείς εκ των υστέρων, χωρίς δικαιολόγηση, χωρίς ε, ε, εξήγηση, χωρίς τίποτα, ότι εντάξει μωρέ, με βόλευε να βάλω μεταλλικές και έβαλα. Ε, αυτό παραβιάζει τους όρους μιας ε, ε, σύμβασης. Και στο ενοχικό δίκαιο στο αστικό δίκαιο ε, είναι ιερό το συμβόλαιο. Ε, συμφωνώ απολύτως και με την κυρία Μάλετης στο συμπέρασμα που καταλήγει ότι χρειάζεται περισσότερη πρόληψη και περισσότερη εκπαίδευση, βεβαίως. Ωστόσο, όταν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιες συμφωνίες μεταξύ των μερών, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ε, νομίζω είναι σαφές αυτό. Ένα τελευταίο. Επανέρχομαι στον εντοπισμό ή την ανείχνευση. Γενικά, είπαμε είναι καλό να αυξάνονται οι αναφορές, είναι θετικό γιατί μπορούν έτσι να διορθώνονται. Αλλά, βεβαίως, οι παρατυπίες που αναφέρονται προέρχονται από διάφορε πηγές ανείχνευση. Δηλαδή, η βασική πηγή είναι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν τα κράτη-μέλη και είναι πάρα πολύ καλό αυτό γιατί σημαίνει ότι δουλεύουν σωστά τα συστήματα, κάνουν τη δουλειά τους και ανοιχνεύουν παρατυπίες και μάλιστα όλες τις παρατυπίες που έχουν γίνει. Μετά τη σύναψη της σύμβασης και κατά τη διάφορα της εκτέλεσής τους από επιτόπιους ελέγχους, από ελέγχους ε, των τιμολογίων, λογιστικούς, ε, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Παρατυπίες μπορούν επίσης να εντοπιστούν από τις ε, αρχές οικονομικού και λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών που έρχονται να ελέγξουν τη διαχειριστική αρχή. Ελεγκτικά συνέδρια, ας πούμε, κλπ. Και μετά υπάρχουν και παρατυπίες που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους ελέγχους της ή το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, η Όλαφ ή ε, από την αστυνομία, τη δικαιοσύνη κτλ. Όλα αυτά τα επίπεδα ελέγχων διαφέρουν. Ορισμένα είναι συστηματικά, είναι εντός του συστήματος, αλλά είναι εξωτερικά. Όταν βρίσκουν κάποιες περιπτώσεις, μας δείχνουν απλώς τη δέσμευση που έχουν και οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές αρχές να ελέγχουν πώς δαπανώνται τα χρήματα και αν είναι σωστή και χρηστή διαχείριση. Αν ήμασταν σίγουροι ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν το ίδιο επίπεδο προσοχής, ας πούμε, όλες οι περιφερειακές αρχές κάνουν τους ίδιους ελέγχους με την ίδια ποιότητα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες παρατυπίες σε μια χώρα δείχνουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι σε άλλα. Σε κάποιο βαθμό αυτό γίνεται με τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο. Δουλειά τους είναι να καταδεικνύουν τα προβλήματα στο σύστημα του ελέγχου, της διαχείρισης και του οικονομικού ελέγχου των Αλλά αν τα δούμε από πλευρά καταπολέμησης απάτης, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη με αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ και πάλι και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας πάντα και παραμένω και του εισηγητού και της Επιτροπής για οποιασδήποτε διευκρινής χρειάζεται περαιτέρω ή ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you for your Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, κυρία Ρημόν, θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσους τους συναδέλφους, όσους από τους συναδέλφους συμμετείχαν στην συζήτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέροντες παρατηρήσεις άκουσα. Θέλω να αναφερθώ σε πέντε σημεία. Μιλήσατε για πραγματικές παρατυπίες, για διάφορες κατηγορίες παρατυπιών. Ναι, βέβαια, μπορούμε να συζητήσουμε για τις κατηγορίες παρατυπιών. Είναι θέμα ορισμού όμως πάλι. Εδώ η έκθεση ουσιαστικά πάσχει από το γεγονός ότι σε πολλά σημαντικά σημεία δεν έχουμε ενιαίους ορισμούς. Δεν έχουμε κοινά αποδεκτά αποδεκτούς ορισμούς και αυτό σε πολλά σημεία επαναλαμβάνω. Δεν έχει νόημα τώρα να μιλήσουμε για μια τεχνική παρατυπία ή μια ουσιαστική παρατυπία. Πρέπει να υπάρξει ενιαίος ορισμός και επαναλαμβάνω ότι στον κανονισμό του 2012-363 η Επιτροπή προσπαθεί να φτάσει σε έναν ενιαίο ορισμό της απάτης. Άμα δείτε το κείμενο είναι αρκετά μεγάλο εξάλλου. Ε, το θέμα είναι βέβαια ότι η απάτη είναι κάτι που αποτελεί μια εσκεμμένη πράξη, ένα αδίκημα, ε, κάτι που περιλαμβάνει ο ποινικό κώδικας όλων των κρατών μελών. Είναι ίσως πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται να φτάσουμε σε μια ε, ενιαία περιγραφή και ενιαίο ορισμό. Το θέμα της παρατυπίας είναι πιο δύσκολο. Το θέμα τώρα του εάν τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για τον σωστό σκοπό. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το επεξεργαστούμε, να το συζητήσουμε. Το θέμα δεν είναι αν τα χρήματα αυτά δόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ε, για, με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά αν δόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες και σύμφωνα με τον αρχικά προβλεπόμενο σκοπό είναι κάτι διαφορετικό και εδώ βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ βασίστηκα πάντα στα κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το θέμα είναι για το θέμα του εισαγγελέα, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, να βασιστούμε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις από μέρους των κρατών μελών. Ε, το θέμα του συντονισμού, το θέμα της δράσης και της Όλαφ, αλλά και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καλαπολέμηση της Απάτης, αλλά και αυτού του νέου ε, γενικού εισαγγελέα, του νέου θεσμού, οι αρμοδιότητες θα πρέπει να καθοριστούν, κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Αναφερθήκατε επίσης πολλοί από εσάς σε περιπτώσεις συγκεκριμένες ε, απάτες. Η Επιτροπή έχει αναφέρει τον εντοπισμό, τους διαφορετικούς τρόπους εντοπισμού και ανείχνευσης κάποιων περιπτώσεων απάτης από τα 28 κράτη-μέλη στα 6 από αυτά τα 28 για το 2013 δεν υπήρξε απολύτως καμία απάτη. Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε γίνονται όλα τόσο ωραία και κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο έτσι ώστε να μην υπάρχει πραγματικά καμία απάτη. Είτε είναι θέμα εντοπισμού ελέγχων και επιπτώσεων για τα κράτη-μέλη τελικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει ότι τίποτα το παράτυπο δεν συνέβη σε αυτά τα κράτη-μέλη το 2013 ή ότι απλώς δεν εντοπίστηκαν οι απάτες και οι παρατυπίες. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για μένα. Εκεί που συμφωνώ με όλους όσους αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό είναι το θέμα των παρατυπιών, πώς ορίζονται οι παρατυπίες και το θέμα της απλοποίησης των κανόνων που σίγουρα θα οδηγήσει σε μείωση των περιπτώσεων σφαλμάτων και παρατυπιών. Εδώ οπωσδήποτε πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτό της απλοποίησης και η απλοποίηση των κανόνων αυτή καθεαυτή σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και στην πράξη και στα νομικά κείμενα σε όλα τα κράτη-μέλη. έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις προσπάθειές μας στις πραγματικές απάντες και στις πραγματικά δόλιες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ όλους πάντως για την συνεισφορά σας. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Αριμόν. Εξαιρετική γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη συνεισφορά και όλους όσοι μίλησαν. Θα μας επιτρέψει αυτό να κάνουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 3 ε, Δεκεμβρίου. Το επόμενο θέμα είναι διάφορα. Έχουμε τίποτα διάφορα. Όχι. Κανένα διάφορο. Επόμενη συνεδρίαση. 3 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη. 9 με 12,5 και 3 με 6,5. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς για την υποστήριξή τους και εμείς ευχαριστούμε. Λήξη της δημόσιας συνεδρίασης ακολουθούν συντονιστές. Παρακαλώ όσοι δεν συμμετέχετε στη συνεδρίαση των συντονιστών να αποχωρήσετε τις αιθούς και να παραμείνουν συντονιστές. Ευχαριστώ.